Let's Ας αρχίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεώς μας. Πάμε στην ακρόασή μας για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης και την καταπολέμηση των λόγων μίσους στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου. Τα θέματά μας είναι πολύ ευραία και ταυτόχρονα διασυνδέονται μεταξύ τους, είναι αλληλένδετα. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην Ευρώπη. Θέλω να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους, να διαφυλάξουμε την εξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, να καταπολεμήσουμε τους ε, λόγους ε, μυσαλλοδοξίας και παραπληροφόρηση επίσης να καταπολεμήσουμε, διότι όλα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δημοκρατία μας. Η δημοκρατία μας, όπως ξέρουμε, βασίζεται στο κράτος δικαίου. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο πλουραλισμός τους και η προστασία των ε, δημοσιογράφων ήταν στο επίκεντρο των, του προγράμματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών έχουμε ένα ρόλο ελέγχου όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Και μέσω των δραστηριοτήτων μας της εποπτείας και του ελέγχου όσον αφορά την που γίνεται εφαρμόζεται από την ομάδα για την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Η ελευθερία και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και ο πλουραλισμός είναι βασικές συνιστώσεις του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης είναι ζωτική σημασία για τη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών μελών αυτή. Παρόλο που πρέπει να επαγρυπνούμε για να διαφυλάξουμε τα θεμελιώδη μας δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, πρέπει να δεχτούμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη υπήρξε μάρτυρας σημαντικής αύξησης λόγων μυσαλλοδοξίας στο διαδίκτυο και εκτός ε, διαδικτύου, σε όλα τα μέσα οι δημοσιογράφοι και άλλοι φορείς των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύουν από πολλαπλές επιθέσεις, απειλές, πιέσεις και δολοφονικές απόπειρες. Ήμασταν μάρτυρες αυτών πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν να υποβάλουμε συγκεκριμένες συστάσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Η παραπληροφόρηση ή η προπαγάνδα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής αυξάνεται. Μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές. Από επίσημους φορείς, από πολιτικούς, από πολιτικά κόμματα, από ιδιωτικούς φορείς, από οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε το πώς θα καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση την εποχή της ψηφιακής μεταμόρφωσης των μέσων ενημέρωσης. Ξεκινάμε με, την με το πρώτο μας θέμα, εστιάζεται στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία των ερευνητικών δημοσιογράφων. Θα ακούσουμε την άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα ακούσουμε την επικεφαλής του Τμήματος ε, Πληροφόρησης και Ελευθερία του κ. Μπένιγκς, ο κ. Πάτρικ Μπένιγκς. Μετά η κυρία Ζούλη Μάιοσακ, επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελών των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Μετά παρουσίαση από πλευράς των ερευνητικών δημοσιογράφων, ο κ. Πέτερ Έρντερλι και ο κ. Νταν Καπολάγκα θα μιλήσουν που εργάζονται στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία αντιστοιχώ. Τα μέλη του πάνελ έχουν ετοιμάσει παρουσιάσεις PowerPoint και ο κ. Ερντελή ζήτησε να διανεμηθεί το υλικό του. Και τώρα να δώσω το λόγο στους φιλοξενούμενούς μας. Ο κύριος Πένιξ πρώτος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, φοβάμαι ότι θα δώσω μια πολύ ζωφερή εικόνα της ε, ελευθεροτυπίας ε, της κατάστασης ελευθεροτυπίας στην Ευρώπη, όχι μόνο στα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και δυστυχώς προσκεκλημένοι μα σίγουρα είναι ότι θα καταλήξουν ε, στα ίδια συμπεράσματα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε κοινέ απαντήσει ε, παρά να παρουσιάζουμε μια ακόμη πιο ζωφερή εικόνα όσο περνάει ο χρόνος. Όλοι συμφωνούμε ότι η ελευθερία των ΜΜΕ είναι πυλώνα των δημοκρατικών κοινωνιών. Αυτό είναι αμφισβήτητο, διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ. Το δυστυχέ είναι ότι πέραν από όλε τι δεσμεύσει μα φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου η ελευθεροτυπία απειλείται όλο ένα και περισσότερο και οι απαντήσεις που δίνουμε δεν είναι και απαραίτητα θετικές συμπεριλαμβανομένων ε, και των ε, κορυφαίων πολιτικών. Να απευθύνω έκκληση λοιπόν ότι κάποια στιγμή μετά την ακρόαση θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ελαφρώς ε, αυτή την εικόνα. Είμαι επικεφαλής ε, του τμήματος ε, της ε, κοινωνίας της ενημέρωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ασχολούμαστε με την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης. Η ελευθεροτυπία δεν αποτελεί μόνο πυλώνα των δημοκρατικών κοινωνιών, αποτελεί ένα δικαίωμα που ρητά καταγράφεται στο Ευρωπαϊκό Συντάγμα για την Προστασία των, Ευρωπαϊκών, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα της διαφάνειας. Θα ήθελα να δούμε κάποιες ε, διαφάνειες. Ε, δεν ε, μπορώ παρά να αναφέρω την υπόθεση της Δέφνα Καρουάνα Γκαλίτσια. Εδώ ακούσαμε στο Στρασβούργο τη συγκεκριμένη κατάσταση, όμως βλέπουμε με σαφήνεια τι συνέβη και τι κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε μια πλατφόρμα για την προστασία των δημοσιογράφων και άλλων ε, απασχολούμενο στα μέσα και λαμβάνουμε ενημέρωση από τους δημοσιογράφους ε, προκειμένου να μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει. Αυτό μας δίνει ένα δικαίωμα να θέτουμε ερωτήσεις στις κυβερνήσεις και να ακούσουμε την αντίδρασή τους. Δυστυχώς δεν υπάρχει το απαραίτητο follow-up σε κάθε περίπτωση και ακόμη και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, έχει ζητήσει να λάβει χώρα ανεξάρτητη έρευνα. Τα νεότερα ήταν ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει θετικές απαντήσεις παρόλη τη δέσμευση των μελτιζικών αρχών να μας απαντήσουν και να κάνουν κάτι τέτοιο. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση λοιπόν είναι το αδελφό όργανο το δικό σας. Τώρα, ποιες είναι οι κυρίες προκλήσεις, ε, τι αντιμετωπίζουμε το 2019. Ε, είδαμε ότι είχαμε δύο δολοφονίες ε, δημοσιογράφων στην Ευρώπη που ερευνούσαν το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφορά. Περιοριστική νομοθεσία όλο ένα και περισσότερο που ουσιαστικά έχει αντίκτυπο ε, στην ε, δυνατότητα να επιβιώσουν οι ποιοτικοί δημοσιογράφοι. Έχουμε διώξεις, ποινικέ ε, διώξεις δημοσιογράφων, όλο ένα και αυξανόμενες ευθύνες των μεγάλων online πλατφόρμων για την διάδοση παραπληροφόρησης και τρομοκρατικής προπαγάνδας ταυτόχρονα ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών και άλλα συμφέροντα. Αυτές είναι προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτή τη στιγμή Υπάρχει περαιτέρω εκφοβισμό, αλλά όχι μόνο εκφοβισμός των δημοσιογράφων, υβριδικέ επιθέσεις και παραπληροφόρηση, ξένη παρέμβαση στις εκλογές, ε, ε, ε λόγο μίσου, ρητορική μίσου, και μιλάμε για το κίνδυνο, για την ελευθερία των ΜΜΕ, ε, κίνδυνος κατά της ελευθερίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων και του συστήματος δημοκρατικής διακυβέρνησης. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε διάφορους τομείς και να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένα στον τομέα της ασφάλειας των δημοσιογράφων, της ελευθεροτυπίας, της ελευθερίας έκφρασης και της ανάπτυξης πολιτικής. Όμως, πολύ συχνά, μόνο η ανάπτυξη πολιτικής δεν αρκεί. Θα πρέπει να μπορούμε να θεσπίσουμε μηχανισμούς που να απαντούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις που σας ανέφερα. Ε, για τον επιγραμμικό, για την επιγραμμική ρητορική μίσους, αυτό είναι μέρος αυτού και θα ε, τα αναφέρω αυτά. Θα τα αναφέρουμε αυτά στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Ένα από τα στοιχεία που σας ανέφερα, και εδώ βλέπετε και τις φωτογραφίες των δημοσιογράφων που πρόσφατα δολοφονήθηκαν, έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο που είναι η online πλατφόρμα για την προστασία των δημοσιογράφων. Ως ε, διακυβερνητικός οργανισμός ε, προσπαθούμε να το προωθήσουμε γιατί είναι ένα από τα στοιχεία που οι εταίροι οργανώσεις δημοσιογράφων ε, μπορούν να συμμετέχουν και να μας ειδοποιήσουν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες αντιδράσεις. Πέραν αυτών, ε, δεν σημαίνει ότι βελτιώνεται η κατάσταση, θα έλεγα το αντίθετο μάλιστα. Φυσικά, εστιαζόμαστε καταρχήν στην προστασία των δημοσιογράφων και μία από τις ε, κύριες συστάσεις εδώ που εκδόθηκε από την ε, Επιτροπή των Υπουργών των 47 κρατών μελών αφορά την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τη δημοσιογραφία, αλλά ταυτόχρονα ε, και ε, να ασκούμε δίωξη αν χρειαστεί σε όσους επιτίθενται στην ελευθεροτυπία. Θα πρέπει να τα θέσουμε όλα αυτά στην πράξη. Θα πρέπει να τα κάνουμε πράξη, να διασφαλίσουμε ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο στα χαρτιά, αλλά υπάρχει και ανάλογη πρακτική στα κράτη-μέλη μας. Επίσης, προφανώς, ε, ο πλουραλισμός των ΜΜΕ και η προστασία των δημοσιογράφων συμβαδίζει με την αυξανόμενη παραπληροφόρηση υπό το φως ε, της επικοινωνίας ε, σε σχέση με τις εκλογές, αλλά και ευρύτερα στην πολιτική ζωή. Εδώ προστίθεται και η απειλή κατά αυτών που θέλουν να δείξουν ε, κάποιες στρεβλώσεις που υπάρχουν στα κυβερνητικά συστήματα. Οι προκλήσεις για το μέλλον. Φυσικά έχουμε αδύναμες ε, νομοθεσίες, ε, έχουμε τα προβλήματα με την ενημέρωση μέσων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ε, και πρέπει να έχουμε και ποιοτική δημοσιογραφία. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, οργανώνουμε και μια σχετική διάσκεψη. Η ανάγκη οι πλατφόρμες στο διαδίκτυο να μπορούν και αυτές να συμβάλλουν για να διασφαλίσουν ότι η ποιοτική δημοσιογραφία πρέπει να προστατευτεί και να προωθηθεί. Και αυτό συμβαδίζει με όλα τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε σε επίπεδο των ενδιάμεσων ε, στο διαδίκτυο. Επίσης, ε, σε επίπεδο κοινοβουλευτική συνέλευση, υλοποιούμε μια σειρά εκθέσεων για το θέμα της ε, ελευθεροτυπίας ε, για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα θεσμό διαμεσολαβητή για τα ΜΜΕ. Επίση, ε, εκπαίδευση, αλφαβητισμό στα μίντια θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους τρόπους δημόσιας συζήτηση, να αποτρέψουμε την εισαγωγή διακρίσεων και επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε δημοκρατική διακυβέρνηση αυτών των νέων εξελίξεων. Βάσει αυτών, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστω να σας απαντήσω κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πένιγκς. Ε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά, κυρία Μαζεζάκ. Καλημέρα σε όλους σας και όλες. Αφού έχουμε διερμηνείς, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα που είναι τα γαλλικά. Euh, Εκπροσωπώ τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα στη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ και 3,5 χρόνια τώρα και όταν άρχισα να δουλεύω για τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και έλεγα που δούλευα μου απαντούσαν συχνά «Α ναι, μπράβο, ωραία, και τι κάνεις ακριβώς εκεί» και αισθανόμουν σε αυτή την ερώτηση μια επιφυλακτικότητα, ένα σκεπτικισμό κατά πόσο χρειάζεται αυτή η δουλειά και ε, η υπεράσπιση, η δημοσιογραφία και η ελευθεροτυπία στην Ευρώπη. Έκτοτε είχαμε το Brexit, το δημοψήφισμα, την εκλογή του Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείες που συχνά αποκαλεί εχθρούς του λαού ε, ε, τους δημοσιογράφους. Μετά είχαμε τη δολοφονία της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίζια, ε, του Γιάν Κούσιακ στη Σλοβακία, μετά τη Μάλτα. Και οι δύο ε, δολοφονήθηκαν επειδή ε, διερευνούσαν θέματα διαφθοράς. Και σήμερα όταν λέω ότι εργάζομαι για τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα μου λένε «Ω, πω, πω, θα πνίγεσαι στη δουλειά και πραγματικά σας έχουμε ανάγκη». Τώρα δεν ξέρω εάν πραγματικά αυτό θα πρέπει να με χαροποιεί αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι η ελευθεροτυπία ταλαιπωρείται, δοκιμάζεται και ότι οι δημοσιογράφοι και ο τύπος ε, διέρχονται μια κρίση εμπιστοσύνης που απειλεί τη δημοκρατία μας. Και η σημερινή ακρόαση είναι εύλογο ως απόδειξη. Ε, θα ήθελα να αρχίσω από τις δολοφονίες των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, που είναι το πιο χαρακτηριστικό. Τρεις δημοσιογράφοι μέσα σε ένα χρόνο δολοφονήθηκαν. 16 Οκτωβρίου 2017 δολοφονείται η Δάφνη Καρουάνα Γαλήσια. Είχαν βάλει βόμβα στο αυτοκίνητό τη στη Μάλτα. Τέσσερι μήνες αργότερα στη Σλοβακία άλλος δημοσιογράφος, ο Γιάν Κούσιακ, 27 ετών, δολοφονήθηκε με πυροβολισμό μαζί με την ε, ε, αρμονιαστικιά του στο σπίτι του και οι δύο δολοφονήθηκαν εσκεμμένα γιατί διερευνούσαν υψηλού επίπεδου διαφθορά. Στις 6 Οκτωβρίου 2018, άλλη δημοσιογράφος στη Βουλγαρία, η Βικτόρια Μαρίνοβα, ε, ε, βιάστηκε βάναυσα και δολοφονήθηκε σε ένα πάρκο στη Βουλγαρία το κίνητρο ακόμα του φόνου αυτού, της δολοφονίας, δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά είχε παρουσιάσει η Μαρίνοβα ε, μία ε, τηλεοπτική εκπομπή για πιθανή διαφθορά με ευρωπαϊκά κονδύλια. Και θέλω να προσθέσω ε, ότι παρατρίχα γλίτωσε από μια τέταρτη δολοφονία δημοσιογράφος στην Ιταλία, χάρη στην αστυνομία αποσοβήθηκε η δολοφονία του ε, δημοσιογράφου από τη Σικελία, Πάολο Μπαρομέτη, ε, ο οποίος ειδικεύεται σε εγκληματικά δίκτυα. Και όταν πιάσανε ένα μαφιόζο σχετικά με την υπόθεση, δήλωσε ότι ε, ένας μικρός θάνατος δρά προειδοποιητικά για τους υπολείπους. Ε, μάλλον τη Ρωσία του Πούτιν θυμίζει αυτή η κατάσταση και λιγότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει. Δυστυχώ, αυτές οι δολοφονίε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου γιατί σήμερα οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι ε, υφίστανται εκφοβισμό και πιέσεις, ε, επιθέσεις, φραστικέ, σωματικέ. Ε, και όλο και περισσότερο δικαστικέ. Όταν συμβαίνει αυτό η δημοκρατία απειλείται. Στην Ιταλία ο Ρομπέρτο Σαβιάνο, ο Πάολο Μπορρομέτη και καμιά εικοσιαριά δημοσιογράφοι ζουν 24 ώρες το 24ωρο υπό αστυνομική προστασία. Αυτή η ανάγκη αστυνομικής προστασίας φαίνεται και σε άλλες χώρες που είναι ε, υποτίθεται ε, στην κορυφή της ελευθεροτυπίας. Στις κάτω χώρες δύο ε, δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στις εγκληματικές οργανώσεις ενοχλούν οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι γιατί διερευνούν τη διεθνή επιρροή και τη διαπλοκή μαφιόζων με πολιτικών για ευρωπαϊκά κονδύλια που χάνονται. Ειδικά στην ε, Βουλγαρία που είναι ουραγός ε, στην ευρωπαϊκή κατάταξη ελευθεροτυπίας. Είναι μια χώρα ε, όπου συχνά στιγματίζεται για την ε, διαφθορά, για τη δικαιοσύνη που είναι αναποτελεσματική και είναι σε μια μέγενη δημοσιογράφη από τη μια το οργανωμένο έγκλημα και από την άλλη ε, η οργανωμένη εξουσία που δεν τους υπερασπίζεται. Παντού, σε όλη την Ήπειρο, όταν υψώνουν τη φωνή τους οι δημοσιογράφοι για κάποια σκάνδαλα που ενοχλούν, τους ψάχνουν δικαστικά και, στη, και τους ενοχλούν και στη Ρουμανία και στην Πολωνία. Ο Τόμας Πιέτεκ ε, από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και τον κατηγόρησαν για τρομοκρατία γιατί είπε ότι ο Πολωνός ε, Υπουργός ε, Αμήνης συνδέεται με τη Ρώσικη μαφία. Ε, και ε, τώρα η εργαζόμενοι στην καζέτα Βιπόρσκα, επίσης διώκονται γιατί αμφισβήτησαν τον Κασίσκι, ε, τον ηγέτη της χώρας που ενέχεται σε περίεργα ε, σχέδια ε, κατασκευαστικά και οικοδομών. Βλέπουμε μια πρακτική αποτρεπτική είναι αυτό που ονομάζεται SLAP στα ε, αγγλικά, ότι στρατηγικά ε, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ε, κατά της δημόσιας συμμετοχής. Αυτό που θέλουν είναι να φημώσουν τους δημοσιογράφους και όχι τόσο πολύ να πάρουν αποζημίωση χρηματική. Θέλουν να τους αφεμάξουν. Και στη Μάλτα το έκαναν αυτό στην Δάφνε Καρουάνα Γαλίτσια και τώρα το χρησιμοποιούν κατά ε, των δημοσιογράφων που είναι μια χούφτα όπως είναι η Καρολίν Μουσκά που προσπαθεί να δώσει συνέχεια σε αυτή τη δουλειά της Δάφνης και που ε, καταδεικνύει ε, το ξέπλυμα χρήματος στο αρχιπέλαγος της Μάλτας. Η Δάφνη υπέστη ε, ε, ε, πραγματικά δικαστική παρενόχληση όταν τη σκότωσαν. Είχε 50 δίκες, συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της. Και σήμερα συνεχίζονται, παρόλο που έχει σκοτωθεί η γυναίκα, 26 μηνύσεις και αγωγές και βαραίνουν τους γιους της. Στη Γαλλία το είδαμε αυτό με το Βενσάν Μπολορέ που μόλις ένας δημοσιογράφος αναφερθεί ε, στις δράσεις του ε, αμέσως ε, προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Στην Κροατία η αντίστοιχη e ΕΣΥΕΑ βρήκε πάνω από χίλιες αγωγές κατά δημοσιογράφων. άλλη απειλή, πολύ σοβαρή, είναι η παρενόχληση στο διαδίκτυο από στρατιές τρόλ που μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα ή μισθοφόροι που τους πληρώνουν αυταρχικά κράτη. Και αυτή η παρενόχληση είναι ένα μέσο εκφοβισμού και ε, φήμωσης των δημοσιογράφων. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει αν δεν το έχει ζήσει, αλλά είναι πάρα πολύ βίαιο και ομό και για να αντισταθεί κανείς θα πρέπει να έχει μια καταπληκτική έτσι, δύναμη και θάρρος και απίστευτη στις 14 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Dark Place και ε, εκεί οι γυναίκες ε, δημοσιογράφοι ε, μαρτυρούν που γυναίκες καταθέτουν τη μαρτυρία τους που έχουν υποστεί τέτοια μορφή παρενόχλησης. Ο ΑΣΕ είναι ο παραγωγός αυτού του ντοκιμαντέρ και ε, πραγματικά η εικονική πραγματικότητα δεν είναι καθόλου εικονική, έχει πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις. Τώρα θα ήθελα σύντομα να πω δύο λόγια για μια άλλη τάση πάρα πολύ ανησυχητική σε πολλές ε, δημοκρατίες που είναι η ρητορική κατά του τύπου. Υπάρχει ένα ε, κλίμα εχθρικό έως και μίσους κατά των δημοσιογράφων στις δημοκρατίες μας. Και αυτό είναι πολύ πιο ανησυχητικό τη στιγμή που ενισχύεται και ενθαρρύνεται από κάποιους ε, πολιτικούς ηγέτες. Όλο και περισσότεροι πολιτικοί ε, δεν θεωρούν τον τύπο ε, θεμέλιο απαραίτητο της δημοκρατίας, αλλά αντίπαλό τους και δεν διστάζουν να του επιτεθούν. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, είναι οι δημοσιογράφοι ανεπιθύμητα πρόσωπα Ούτε ο Όρμπαν τους μιλάει, αν δεν είναι ε, από μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν το Φιντές. Στη Γαλλία, ε, ο Μελανσόν ε, της ανυπότακτης Γαλλίας γράφει στο blog του. Το μίσος για τον τύπο είναι υγιές και σωστό. Τον Οκτώβριο του 2017 συνέβη κάτι τρομακτικό και θέλω να το θυμίσω. Ο Τσέχος πρόεδρος Μίλος Ζέμαν ήρθε σε συνέντευξη τύπου με ε, ένα πλαστό καλάσνικοφ και πάνω έγραφε για τους δημοσιογράφους. Το έχω φέρει το καλάσνικοφ αυτό. Αυτές οι φραστικές επιθέσεις και οι απειλές δεν είναι απλώς δυσάρεστες, είναι επικίνδυνες. Δηλαδή ε, καλούν ε, στο, στη σωματική βία. Το είδαμε στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, άνευ προηγουμένου βία. Ε, ορισμένες τηλεοράσεις ε, δεν μπορούν να κατέβουν με κάμερες που να γράφουν το κανάλι ή να στέλνουν δημοσιογράφους χωρίς να συνοδεύονται από σωματοφύλοκες για την προστασία αυτών των ερευνητικών δημοσιογράφων θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία και ελευθερία. Σε πολλές χώρες όμως οι ολιγάρχες χτίζουν ή αγοράζουν ολόκληρες αυτοκρατορίες. Αγοράζουν ε, τα μίντια όχι για να αυξηθεί η πολυφωνία, αλλά για να την υποτάξουν ε, στην οικονομική τους η πολιτική εξουσία. Ε, οι τράπεζες, τα τηλέφωνα, η οικοδομή, τα δημόσια έργα, ε, συνδέονται με διαπλοκή σύγκρουση συμφερόντων και στρέφονται κατά των δημοσιογράφων και κατά του δικαιώματος του καθενός να έχει ε, ε, μια τίμη ενημέρωση στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία, στη Τσεχική Δημοκρατία. Και για να είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα, έχουμε τώρα και την παραπληροφόρηση. Ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης είναι ότι ε, στερεί αξιοπιστία από όλη την επικοινωνία. Τα fake news ε, καταρρύπτουν και τις σωστές πληροφορίες των ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Σήμερα ο κόσμος σου λέει «Α, το διάβασα στο Facebook». Το διάβασα στο Facebook δεν ξέρουν πια τι είναι τύπος, τι είναι μέσα ενημέρωσης, τι είναι γεγονός, τι είναι αξιόπιστη πηγή, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Δεν υπάρχουν πια αλήθειες, δεν υπάρχουν γεγονότα. Υπάρχουν μόνο απόψεις, εναλλακτικά γεγονότα, ε, συναισθήματα. Ε, ακόμα και το Russia Today έχει φτιάξει fact-checking, μια επιτροπή για να ελέγχει τα γεγονότα. Ε, χρειαζόμαστε ανεξάρτητη, λοιπόν, ε, ε, ανεξάρτητο τύπο και μίντια στην Ευρώπη που να ενημερώνουν τους πολίτες να καταγγέλουν τις καταχρήσεις. Αν δεν είναι ελεύθερος ο τύπος, δεν ακούγεται κανένας αγώνας πουθενά. Και προς τα εκεί ολισθαίνουν τα καθεστώτα προς την ολοκληρωτική ε, τακτική. Φημώνουν τον τύπο. Αυτό που χρειάζεται είναι ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, αυστηρά, σοβαρά. Μεγάλη πρόκληση. Κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ, η ρεπόρτερ χωρίς σύνορα κάναμε 10 προτάσεις για να προστατεύετε καλύτερα ελευθεροτυπία στην Ευρώπη. Σας έχω φέρει εδώ κάποια αντίτυπα, αν σας ενδιαφέρει. Ε, επειδή πρέπει να τελειώσω, ήθελα να μιλήσω για κάποιες από τις προτάσεις αυτές πάρα πολύ σύντομα. Πρώτον, να υπάρχει ένα σύνδεσμος ε, έκτακτης ανάγκης, ε, έτσι ώστε επιγόντως να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Ε, ένα σημείο επαφής που θα μπορούσε να είναι επίτροπος που θα μπορούσε να δρά σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές για να προστατεύεται η ελευθερία της ενημέρωσης. Επίσης, μέτρα κατά του ΣΛΑΠ αυτής της δικαστικής παρενόχλησης. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στην κατάσταση της ελευθερίας του τύπου. Οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάζει περιοδικά την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου σε όλα τα κράτη-μέλη και να καταλήγει σε συστάσεις ενδεχομένως ανά χώρα και σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις να προβαίνει και σε κυρώσεις. Δηλαδή να σταματούν ε, οι χορηγήσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων στις εν λόγω χώρες. Και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έργη, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, είμαι ο Πίτο Ρέτη και είμαι δημοσιογράφος και εκδότης στο, στον Ουγγρικό τύπο. Έχουμε περίπου 400.000 επισκέπτες την ημέρα. Καλύπτουμε δημόσια θέματα και έχουμε κερδίσει πολλά βραβεία για τον ερευνητικό μας, ε, το ερευνητικό μας έργο. Έχουμε λοιπόν αυτή την πύλη για τις ειδήσει. Λοιπόν, αριστερά βλέπετε το, τα γραφεία του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας που εργάζονται οι βουλευτές. Στο ισόγειο βλέπετε κάτω με, με το κομμάτι αυτό που είναι 10 τετραγωνικά μέτρα. Πρόσφατα το προσθέσανε. Ο πρόεδρο τη Βουλή καθόρισε ότι αυτό είναι ο χώρο δημοσιογράφου. Παρόμοιο χώρο ε, είναι και στο Κοινοβούλιο. Οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν σε, και να παίρνουν συνέντευξη από τους βουλευτές εκτός του Κοινοβουλίου. Όταν ρωτήσεις, ε, ρωτήσεις εκτός του Κοινοβουλίου, αυτό έχει ειδικά του προβλήματα που δημιουργούνται. Ένας βουλευτής, ε, ε, ένας βουλευτής του ΦΙΝΤΕΣ ε, ε, εμείνει σε ένα δημοσιογράφο για παρενόχληση όταν θέλεις να του ρωτήσεις. Όταν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι πήγαν στην πατρίδα του Ορμπάν να πάρουν ε, συνέντευξη, τους έψαξαν οι αστυνομικοί, ζήτησαν ταυτότητες κλπ. Ε, και, και, είχαμε και κάποιες κατασχέσεις ε, των μηχανημάτων. Το ψηφιακό μονοπάτι είναι πιο εύκολο. Email που στέλνετε στου πολιτικού, του φίδε και αξιωματούχου και θεσμού ε, πάντα αγνοούνται σχεδόν. Ο Πρωθυπουργό Ορμπάν δεν έδωσε συνέντευξη σαν εξάρτητο ε, δημοσιογράφο πάνω από, εδώ και πάνω από πέντε χρόνια. Λοιπόν, πριν ανέβει το 2010 το Φίντε στην εξουσία, είχαμε πολύ προοδευτικού νόμου στην Ουγγαρία, στην Ευρώπη χρησιμοποιούσαν λοιπόν τα αίτημα για να αποκαλύψουν τη διαφθορά οι δημοσιογράφοι. Άλλαξε ο νόμο. Οπότε οι κρατικοί θεσμοί μπορούν χιλιάδε ευρώ να επιβάλλουν, να ζητήσουν για να μπορέσουν να απαντήσουν θετικά σε αίτημα. Το Νότο Δικαστήριο αποφάσισε πρόσφατα ότι ο, ο, του Πρωθυπουργού Ορμπάν, ο οποίο παίρνει πολλού πόρου ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δημόσιο πρόσωπο. Ο Τίμπος, και ο δημοσιογράφος τους, ο δικηγόρος τους ζήτησε να μην τον ενοχλούν άλλο. Και έγινε, δηλαδή, τελικά η νομοθεσία τους καλύψαν ιδιωτικά πρόσωπα, από που δημόσια πρόσωπα. Λοιπόν, όταν οι δημοσιογράφοι τους ρωτάνε ερωτήσεις, θεωρείται ότι παρεμβαίνουν στην ιδιωτική του ζωή και τους παρενοχλούν. Ανεξάρτητη δημοσιογραφία απειλείται. Έχουμε δημοσίευση τη άκρα δεξιάς που αφορά, αναφέρεται στη, δεξιά μου, στην δική μου ε, εφημερίδα και λένε είσαστε ε, οι μεγαλύτεροι εχθροί των Ούγγρων και θα πρέπει να σας εξαλείψουμε από την ε, Ουγγαρία. Ότι είστε ακροδεξιοί και εξτρεμιστές. Κάθε χώρα έχει βίου εξτρεμιστές. Ποια είναι διαφορά στην Ουγγαρία. Ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου και Κυβέρνηση χρησιμοποιούν τις σελίδες τους του Facebook για να ποστάρουν θέματα από αυτό το αυτήν την εξτρεμιστική ιστοσελίδα. Παρουσιάζεται ε, επίσης δεν πηγαίνουν κατά εκφράσεων ακραίων και απειλούν οι αρχές και παρενοχλούν. Ένας δημοσιογράφος, συνάδελφος, προσεγγίστηκε από τη μυστική υπηρεσία. Του δείξαν φωτογραφίες από την ιδιωτική του ζωή και του είπαν ότι κοιτάξτε, κάποιο μπορεί να σα εκβιάσει με αυτά. Συνεργαστείτε με την κυβέρνηση για το καλό σα, να σα προστατεύσουμε. Η κίνηση κατά των εξαρτήτων μέσων είναι κίνηση τη ε, κυβέρνηση που έφτιαξε αυτοκρατορία. Πριν από ένα χρόνο, δημοσιογράφοι ιδιοκτήτε από πάνω από 400 μέσα ενημέρωση αποφάσισαν όλο το χαρτοφυλάκιο για τα ΜΜΕ να τα βάλουν στο κεντρικό ίδρυμα για τα μέσα ενημέρωση. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Πρωθυπουργό Ορμπάν υπέγραψε διάταγμα και εξαίρεσε τη συγχώνευση από έλεγχο άνευ κεντρική προσέγγιση όσον αφορά τα ραδιοτηλεπτικά δίκτυα, τον τύπο, τα πάντα. Όλα συγκεντρωτικά σε ένα σημείο, σε, σε ένα φορέα. Δημιουργήθηκε αυτό το ίδρυμα. Μία μέρα πριν από τι εκλογέ στι 26 Μαΐου, αυτέ ήταν οι πρώτε σελίδε από το σελίδα κάθε περιφερειακή εφημερίδα στην Ουγγαρία. Τίτλο. Αναφέρεται στι εκλογέ την επόμενη μέρα και λέει ότι θα πρέ... είπε ο Ορμπάν τότε, θα είναι όλοι που είναι υπέρ τη μετανάστευση να είμαστε κι εμεί εκεί. Έμεσα χρηματοδοτεί φορολογούμενο όλα αυτά. Η Ένωση Διαφημιστών τη Ουγγαρία αναφέρει ότι το κράτο είναι ο μεγαλύτερο διαφημιστή στην Ουγγαρία. Δεν είναι αυτοκινητοβιομηχανία ούτε οι τράπεζε. Η κυβέρνηση κάνει εκστρατείε για τα κακά που κάνουν οι Βρυξέλλε, η μετανάστευση κλπ. Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ έχει εξοδεύσει η κυβέρνηση διαφημίζοντα όλα αυτά. Αποκριστικά, διαφημίζουν μέσω φιλοκυβερνητικών πηγών και μέσων. Αριστερά τι βλέπετε, το, την ακροματικότητα των μεγαλύτερων καναλιών στην Ουγγαρία. Το TV2 στα κόκκινα που είναι φιλοκυβερνητικά και το RTL που είναι γαλάζιο, που επικρίνει κάπως το καθεστώς δίπλα είναι όσον αφορά την ε, θεαματικότητα. Δεξιά βλέπετε το ποσοστό κρατικών διαφημίσεων. Δεν είναι δύσκολο να πει κανεί ποιο κανάλι το στηρίζει η κυβέρνηση μέσω διαφημίσεων. Οι ιδιωτικέ εταιρείε επίση προσέχουν που διαφημίζουν. Δεν θέλουν να ταράξουν την κυβέρνηση. Και έτσι τα ανεξάρτητα μέσα φυτοζωούν. Ο προπολογισμό του 2020 για τα δημόσιου σταθμού τη Ουγγαρία, όπω αποκαλούνται, τα κρατικά μέσα, θα πω έτσι, έχουν κονδύλι 232 εκατομμύρια ευρώ για τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με πρώην δημοσιογράφο του σταθμού που παρετήθηκε λόγω παρέμβασης της χώρας, υπάρχουν σαφείς οδηγίες να δείχνουν αρνητικά την αντιπολίτευση στα κανάλια. Κατά τις εκλογές, οι κρατικοί σταθμοί πέντε λεπτά δίνουν σε κάθε κόμμα, αλλά εκτός αυτής της περίοδου οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης δεν βγαίνουν στην οθόνη. Ποτέ δεν καλούνται συνεντεύξεις και σε διάφορα προγράμματα. Το Δεκέμβρη πέρασε, ομάδα των, αντι... των βουλευτών της αντιπολίτευσης πήγαν εκεί στους χώρους του σταθμού για το make-up και λοιπά για να διαμαρτυρηθούν. Κάποιοι τους πέταξαν έξω παρά την ασυλία τους. Και πρόσφατα κέρδισαν την πρώτη τους δίκη κατά του κρατικού σταθμού για αυτό που τους έκαναν. Τα κρατικά μέσα της Ουγγαρίας ε, διοχετεύουν μαζικά τη ρωσική προπαγάνδα. Καλύπτουν εξωτερικέ υποθέσει στο Sputnik και του RT του Russia Today, ε, που είναι τα βασικά φερέφωνα του ρωσικού καθεστώτο. Για το TV2 να σα πω, που είναι φιλοκυβερνητικό σταθμό, που παίρνει πολλά χρήματα. 12 Σεπτέμβρη 2018, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση Σαρτζεντίνη. Το TV2 10 λεπτά αναφέρθηκε σε αυτό το βράδυ στι ειδήσει. Εντάξει, σημαντικέ ειδήσει στην Ουγγαρία. Ο παρουσιαστής ξεκίνησε και λέγοντας στα κοινωνικά μέσα προωθούν τον Όρμπαν. Παρά το ότι υιοθέτησε την έκθεση Σαρτζεντίν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επιτυχία την πήρε ο Ορμπάν. Άκουσαν 12 απόψεις υπέρ της κυβερνήσεως στο πρόγραμμα, υπουργό εξωτερικών, πρωθυπουργό, ευρωβουλευτές του Φίντες και φιλοκυβερνητικούς σχολιαστές. Και η αντιπολίτευση Τίποτα. Τι είπαν, μια φράση για αυτούς. Η αντιπολίτευση, κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευση Ουγγαρία ψήφισαν κατά αυτού. Και υποτίθεται αυτή είναι κατά τη Ουγγαρία. Ο Ιστφαν Χουχέι επέβαλε καταγγελία κατά των αρχών. Διότι τα δημόσια κανάλια είναι αμερόληπτα υποτίθεται. Και είπε ότι αυτή η ημεροληψία ήταν υπερβολική. Το ΦΙΔΕΣ του 2011 δεν συμφώνησε με αυτό, ούτε τα μέσα ενημέρωση, ούτε η αρμόδια Δεν βρήκε ότι υπήρξε μεροληψία. Το δικαστήριο έκανε δεύτερη έρευνα. Ε, ακόμα θεωρήθηκε αμερόληπτη η προσέγγιση. Γιατί τη φορά έκανε ο βουλευτή έφεση και μετά από ένα χρόνο από την εκπομπή, μετά την τρίτη έφεση, αποφασίστηκε ότι η εκπομπή ήταν μεροληπτική, αλλά δεν επιβλήθησαν ε, κυρώσει κατά του σταθμού που μεροληπτούσε υπέρ τη κυβέρνηση. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούνται να απειλούν τους αντιπάλους και να λασπολογούν. Κάποια μαθήτρια έγινε στόχος ε, λασπολογίας γιατί μίλησε κάτι της κυβέρνησης. Κάποιος την αποκάλεσε πόρνη και έδειξε επίσης και φωτογραφίες που είχαν παρθεί από κάτω να φαίνεται σχεδόν κάτω από τη φούστα το πόδι της. Λοιπόν, επίσης παραμορφώνονται οι εικόνες ε, των μελών της αντιπολίτευσης, τους παρουσιάζουν με πιο σκούρο δέρμα. Αυτό για να θεωρεί ε, ο, βλέπετε εδώ πώς αλλάζουν η ποια είναι η αρχική εικόνα και πώς μετά με αλλάζουν και ακόμα και τον τόνο του δέρματος για να έχει αρνητική αντίποση αυτός που διαβάζει. Θα μπορούσα να μιλάω για μέρες αναφέρομαι. Είμαι πολύ λογάς, δεν το κάνω. Πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Αυτά δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν εκπροσωπούν την άκρα δεξιά. Απλώς παραπλανούν τον κόσμο, ε, πουλάνε προπαγάνδα, ελέγχονται από την κυβέρνηση, είναι αποτελεσματικά τα ΜΜΕ αυτά, οπότε χρειάζεται τώρα και εξαγωγή. Οι επιχειρηματίες οι Ούγγροι δημιουργούν στη Σλοβενία και στη Μακεδονία παρόμοιε αυτοκρατορίε. Και ο, και ο Hans Christian ο πρώην καγκελάριο τη Αυστρία, είπε ότι και αυτό θέλει να δει κάτι παρόμοιο στην Αυστρία. Έπρεπε μετά από αυτά να παραιτηθεί. Τέλο αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλέ χώρε στον κόσμο υπάρχουν όπου είναι επικίνδυνο να κάνει δημοσιογράφο. Αλλά αυτά συμβαίνουν εδώ, στην Ουγγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούγεται ξένο. Κάτι που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Σας διαβεβαιώνω ότι μπορεί να συμβεί αυτό και στην πατρίδα σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντελή. Κύριε Ταπαλάγα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Λέγομαι Ντάντα Παλάγα, είμαι ερευνητής δημοσιογράφος και εργάζομαι για το G4 Media. Πρόκειται για ένα μικρό ανεξάρτητο, μια μικρή στο σελίδα που ίδρυσα πέρσι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα. Θα κάνω την παρουσίασή μου στη μητρική μου γλώσσα και θα ξεκινήσω τώρα. Όλα ξεκίνησαν ε, περίπου τρία χρόνια πριν από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι το Μάιο του 2019 όταν ε, καταδικάστηκε σε 3,5 ετικά άθρηξη στο Λίβιο ε, ηγήθηκε της Ρωμανίας, de facto, κατά το στυλ του Βίκτορ Όρμπαν. Άσκησε την εξουσία σαν ε, ένας Όρμπαν ή ένας πιο μικρός Ερντογάν, ε, αλλά λιγότερο επιθετικά. Όταν κέρδισε τις εκλογές πριν τρία χρόνια, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, είχε ήδη τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση με αναστολή για κλοπή ψήφων. Η ρουμανική νομοθεσία απαγορεύει σε κάποιον καταδικαστέντα να γίνει πρωθυπουργό. Συνεπώ, ο Ντράγκνεα δεν μπορούσε απευθεία ε, να και τη Ρουμανία όπω όρταν στην Ουγγαρία, Ερντογκάν στην Τουρκία, ε, αλλά μόνο με άλλου ενδιάμεσου, ε, με πρωθυπουργού μαριονέτε που του κατέβαζε όταν αρνούνταν να πάνε πολύ μακριά στον αγώνα του κατά τη δικαιοσύνη. Ε, άλλαξε τρει ε, πρωθυπουργού σε τρία χρόνια. Ε, η πρώτη προτεραιότητα του Λίβιου Ντράγκνε όταν πήρε την εξουσία ήταν να ξεφύγει από το δεύτερο ποινικό, τη δεύτερη ποινική υπόθεση, όπου τον κατηγορούσαν για πλασματικέ προσλήψει. Ήξερε ότι κινδύνευε να καταδικαστεί σε κάθριξη. Σήμερα ο Ντράγκνα βρίσκεται στη φυλακή, όμως όταν ε, ήταν ελεύθερος έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη. Προσπάθησε να καταστρέψει ολόκληρους ε, ε, θεσμούς, να ελέγξει τους δικαστές, να κάνουν να σιωπάσουν οι δημοσιογράφοι, οι ΜΚΟ, οι πολιτικοί, οι αντίπαλοι στράφηκε κατά των επικριτικών ε, φωνών ε, που αποκάλυψαν ε, την κατάχρηση εξουσίας ή το απειλούσαν την ελευθερία. Αγωνίστηκε κατά όλων που αρνήθηκαν να βλέπουν παθητικά πως ένας άνθρωπος τεινάζει στον αέρα τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαφύγει της φυλακής. Έθεσε τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή πορεία της Ρουμανίας στο μεγαλύτερο κίνδυνο των τελευταίων 30 ετών από την πτώση του κομμουνισμού. Όμως, ε, τι τον σταμάτησε από το να καταστρέψει μεθοδικά μια ολόκληρη χώρα τον ε, εντόπισε μία χούφτα δημοσιογράφων, ε, κάποιοι δικαστές ε, που είχαν θάρρος και από την αντίδραση των ανθρώπων στο δρόμο. Θα σας αναφέρω στη συνέχεια μόνο κάποια επεισόδια, όλα είναι άμεσες προσωπικές εμπειρίες και βασίζονται στη γεγονότα και σε δημόσιες δηλώσεις. Στις αρχές του Ιανουαρίου 2017 μία εμπιστή με ειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ήθελε να ποινικοποιήσει με διάταγμα, έκτακτο διάταγμα μία σειρά ποινικών πράξεων με σκοπό να ξεφύγει από την ποινική υπόθεση ο Ντράγκνεα. Το hotnews.ro έγραψε ε, για την πρόθεση της κυβέρνησης και εξήγησε πώς ε, ο να θέλει να τροποποιήσει το ποινικό κώδικα. Οι αποκαλύψεις του Hot News Raw ε, που δημοσιεύθηκαν ε, και σε άλλα ΜΜΕ έβγαλαν χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο για ολόκληρε εβδομάδες. Δεκάδες χιλιάδες Ρουμάνοι διαμαρτυρήθηκαν ε, στην πλατεία μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο. Καθώς φοβήθηκε από το εύρος των διαδηλώσεων, που ήταν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 1989, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ακυρώσει αυτό το, το διάταγμα το έκτακτο. Ένα άλλο επεισόδιο τώρα. Μετά από κάποιους μήνες, το Μάιο του 2017, δημοσίευσα μία σειρά ερευνών ε, για ένα νησί στο Δούναβι, την Πελίνα, που κατέληξε στην οικογένεια Ντράγκνα στη συνέχεια συνέχεια είχε γίνει το αγαπημένο μέρος ψαρέματο και χαλάρωση για τον κύριο Ντάγνε. Ο μικρός παράδεισο που βρίσκεται στο Δουνεβί στην Νότια Ρουμανία πέρασε από το κράτο ε, στου ιδιώτε με κυβερνητική απόφαση. Η κυρία Πλούμ το βοήθησε ε, σε αυτή τη διαδικασία που προτάθηκε για Ευρωπαία Επίτροπο από ε, τον, την κυρία Βιωρίκα την Πρωθυπουργό Μαριονέτα του κυρίου Ντράγκνεα. Σκεφτείτε λίγο ένας ε, πολιτικός ε, κλέβει ένα μέρος του δυναμή με την βοήθεια της κυβέρνησης και κόβει ένα κομμάτι από τη χώρα του, κόβει ένα νησί μόνο για αυτόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνοιξαν ε, οι ερευνητέ μια έρευνα, αλλά δεν ε, μπόρεσαν ε, να ερευνήσουν την κυρία Πλούμπ, γιατί δεν ήρθε η κοινοβουλευτική ασυλία τη κυρία ε, Πλούμπε Η υποψηφιότητα τη εντωμεταξύ απορρίφθηκε στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λόγω των ε, προβλημάτων ε, ακυρεότητες που είχε στην υπόθεση Μπελίνα. Ε, παράλληλα με τις αποκαλύψεις για τον νησί Μπελίνα, οι συνάδελφοι από το Rice Project έγραψαν το 2017 για τις πολυτελείς διακοπές που ο ηγέτης του ΠΣΔ, κόμματος της αριστεράς, υλοποίησε στην Φορταλέσσα στη Βραζιλία. Ένα μήνα αργότερα, τον Ιούνιο του 2017, οι φορολογικές αρχές ε, έκαναν έλεγχο στο Hot News Bureau και στο Rice Project ε, προκειμένου να εκφοβήσουν αυτά τα μέσα. Ο έλεγχος κράτησε έξι μήνες. Παρενόχλησε εξουσία δύο μικρές ε, συντάξεις γιατί τόλμησαν να γράψουν για το μεγάλο αφεντικό. Συνεχίσαμε όλο αυτό να δημοσιεύουμε ερευνές του κυρίου Ντράγκνε που προσπαθούσε να καταστρέψει τη δικαιοσύνη και τον ποινικό κώδικα μέσω έκτακτων διαταγμάτων. Ακολούθησαν και άλλες αποκαλύψεις ε, για μεγαλύτερες υποθέσεις που ξεπερνούν τα σύνορα, περνούν τα σύνορα της Ρουμανίας. Το Φεβρουάριο του 2018 αποκαλύψαμε σε μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε από το hotnews.ro τις ε, λεπτομέρειες μιας μυστικής συμφωνίας που εγγράφτηκε από μια ε, εταιρεία που της έχει ένας ε, από τους fundraiser του Donald Trump και μιας εταιρεία κρατικής Ρουμανίας που εξειδικεύεται στην παραγωγή οπλισμού. Ο στόχος ήταν να υπάρξει μια σύμβαση ε, αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε εταιρεία. Ο Έλιον Μπρόντε, ο ιδιοκτήτης της, ήταν ο ίδιος που είχε καλέσει το Λίβιο Ντράγνεα όταν στην ορκομοσία του Ντόναλτ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2017. Ο Μπρόιτι σήμερα είναι υποδικαστική έρευνα, καθώς είναι υποπτός ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την επιρροή που είχε από τον πρόεδρο Τραμπ για να διευρύνει τις επιχειρήσεις του στη Ρουμανία. Εν συντομία, ο Ντράγκνα προσπάθησε να κάνει ισχυρού συμμάχου στην Άσικτον και να αγοράσει την ανοχή του, ελπίζοντα ότι θα υπάρξει η διάσωσή του πέρα από τον Ατλαντικό. Ήταν ε, ε, διατεθειμένος να πληρώσει οτιδήποτε, αλλά όχι με δικά του χρήματα. Αυτή η έρευνα ε, επί των ε, άνθρωπο λόμπι του του Τραμπ στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στη Hot News ο Λάιοντ Μπρόντι μας απείλησε με μία πολύ κοστοβόρο δίκη στο Λονδίνο και εγώ ίδιος κλήθηκα να συμμετέχω σε μία δίκη που είναι πάρα πολύ ακριβό να περασπιστείς τον εαυτό σου. Ε, τώρα, ε, αποφασίσαμε ε, μαζί με τον Κριστιαν Παντάζη, τον συντάκτη του Hot News δεν είναι καλό να εκθέτουμε ήδη ένα μέσο μας κατά αυτόν τον τρόπο και έτσι ιδρύσαμε το δικό μας site g4media.ro και βασιστήκαμε κυρίως σε ανεξάρτητη χρηματοδότηση και σε δωρεές. Χωρίς την βοήθεια των πολιτών δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Τον Απρίλιο του 2018 το G4 Media Raw ε, ε, δημοσίευσε λεπτομέρειες για την πρόθεση της κυβέρνησης ε, να υιοθετήσει ένα μνημόνιο με το οποίο η Ρουμανία θα υποστήριζε τη μεταφορά της πρεσβείας από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ ήταν η μόνη κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξε την πολιτική των Ηνωμένων στον τομέα αυτό. Δεν υιοθετήθηκε αυτό το μνημόνιο γιατί αντιτάχθηκε ο πρόεδρος Κλάους Γιωχάνης. Ένα άλλο επεισόδιο λαμβάνει η χώρα στις 9 Μαΐου, την μέρα της Ευρώπης, σε μια επίσημη δεξίωση. Αρνήθηκα να σφίξω το χέρι του Λίβρου Ντράγκε, ο οποίος ήρθε χαροπός να με χαιρετήσει, σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Αυτή τη φορά δεν ε, θα κάνουμε χειραψία, του είπα. Γιατί με ρώτησε. Αφού του εξήγησα ποιοι είναι οι δύο λόγοι, ε, για να μην του σφίξω το χέρι, μου είπε με ένα απειλητικό τόνο, μάλιστα, τότε δεν θα δώσουμε το χέρι μέχρι το τέλος. Μετά από λίγε μέρε, ο Λίβριντ ζήτησε δημόσια να ε, τύχω εισαγγελική έρευνα, ε, γιατί το μνημόνιο αυτό ε, ήταν εμπιστευτικό και ο ίδιο έμαθε από τον τύπο την ύπαρξή του. Την ίδια μέρα αυξήθηκαν σημαντικά οι δωρέ από το κοινό. Έτσι λοιπόν αισθάνθηκα ότι πάλι μα στήριζαν οι αναγνώστε. Το καλοκαίρι του 2018 η κυβέρνηση προσπάθησε να υιοθετήσει ένα έκτατο διάταγμα για να διασώσει τον Τάγνα μέσω της τροποποίησης του ποινικού κώδικα ε, και τι δεν είχε λυθεί το πρόβλημα και περνούσε ο χρόνος. Κάθε φορά που ετοιμαζόταν να υιοθετήσει ένα έκτατο διάταγμα, οι πηγές του G4 Media έκαναν το καθήκον τους ε, και σήμερα τους οφείλουμε πολλά. Υπό συνεχή πίεση της ε, κοινή γνώμης και επεξωτερική πίεση που ασκήθηκε και από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση υπαναχώρησε. Ο Λίβρο Ντράγνε και το κόμμα του κατόρθωσαν όμω να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα και τον νόμο περί δικαιοσύνης και άλλαξαν να καταφέραν να απολύσουν και τη Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεση, την πρώην επικεφαλής της εισαγγελία κατά τη διαφθορά. Σήμερα η κυρία Κέβεση είχε επιλεχθεί ως ε, Ευρωπαϊκή Αγγελέα, παρά που δεν την υποστήριξε η κυβέρνησή της. Με συγχωρείτε που μακρηγορώ, χρειάζομαι ακόμα ένα-δύο λεπτά μια, ένα ειδικό ε, τμήμα ε, έρευνας ε, των εισαγγελέων προσπάθησε να παρεμποδίσει την Λάουρα Κοντουρτσοκέβεση από το να αναλάβει επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και τώρα ένα πιο δραματικό επεισόδιο για την Ρουμανική Δημοκρατία. Στις 10 Αυγούστου 2018 η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, άσκησε βία σε μία διαδήλωση που οργανώθηκε στο Βουκουρέστι από τη Ρουμανική Διασπορά που υποστήριζε το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Και πάλι είχαμε επίθεση στην ελευθεροτυπία. Το Νοέμβριο του 2019, συνάδελφοι από το Rights Project δημοσίευσαν μία σειρά γράφων ε, για ε, τις ε, υποθέσεις της συνοδού του Ντράγκνεα στην Βραζιλία και την επόμενη μέρα ζητήθηκε από την αρμόδια αρχή πρόσβαση στα αρχεία μας και μας απείλησαν με πρόστιμο 20 εκατομμυρίων λέει. Ε, και αυτή είναι μια άλλη κατάχρηση του κανονισμού GDPR, προσπάθησαν να μας εκφοβήσουν και πάλι. Όλα ε, σε αυτές οι δράσεις και πολλές άλλες ε, έθεσαν τη Ρουμανία δίπλα στην Ουγγαρία και στην Πολωνία στα πλαίσια ανελεύθερων καθεστώτων που δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Όμως οι πολίτες Ρουμανίας πήραν την εκδίκησή τους στις ευρωπαϊκές εκλογές το Σοσιαλιστικό Κόμμα ε, τιμωρήθηκε στην ψήφο στις 27 Μαΐου. Το Ανώτο Δικαστήριο καταδίκασε το Λίβιο Ντράγκνα σε 3,5 έτη κάθριξης. Αυτές ε, οι φρικτές πράξεις ε, κατά του τύπου, η συνεχής επίθεση κατά της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου έγιναν και πάλι θα σα το λέω, σε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χωρί οι Βρυξέλλες να μπορούν να παρεύουν. Ξέρουμε δεν είναι πολύ καλή κατάσταση ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στην Πολωνία, ούτε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σήμερα η πολιτική κατάσταση της έχει αλλάξει ριζικά. Η κυβέρνηση του ΠΣΕΝΤ έπεσε μετά από πρόταση μορφή τη αντιπολίτευση, Η Βιωρή Καντεμψίλα, η τελευταία μαριονέτα του Ντράγκνα, έφυγε στο Βουκουρέστι. Την Δευτέρα ανέλαβε ναι, νέα κυβέρνηση και τον νέο πρωθυπουργό τον λένε Λούντεβι Κόρμπαν. Θα γελάσετε ελπίζουμε ότι δεν θα θέλει να μιμηθεί το Βίκτορ Όρμπαν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τον ανεξάρτητο είπα και την ελευθερία τη έκφρασης, αλλά ξέρω ότι μπορείτε να μην ε, κάνετε. Παραδείγματο χάρη, μπορείτε να μην θέτετε στα χέρια των πολιτικών ε, νόμου που μπορεί να του χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για να περιορίσει την ελευθερία τη ε, έκφραση. Ο GDPR αποτελεί μόνο ένα, μια άχρηστη νομοθεσία που δεν προστατεύει τους πολίτες περισσότερο από πριν, αλλά σίγουρα κάνει πιο πολύπλοκη τη ζωή των ανεξάρτητων δημοσιογράφων που δεν έχουν πάρα πολλού πόρου Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν μπορούν να σκεφτούν περισσότερο όταν δίνουν ε, στα λόμπι του μεγάλου τύπου ε, τα πάντα και θυσιάζουν τον ανεξάρτητο τύπο. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να προστατεύσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία που είναι πολύ πιο ευάλωτη. Όμως που είναι τα καλά νέα ε, και οι εχθροί της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χάνουν ε, το αγώνα με τους πολίτες. Ε, κάποια στιγμή ε, λάμπει η αλήθεια και φαίνεται στις εκλογές. Και θα κλείσω λέγοντας ότι αυτό το κείμενο το αφιερώνω στους ερευνητές δημοσιογράφους Γιάν Κούτσακ από τη Σλοβακία και την Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσι από τη Μάλτα. Ε, αυτοί κινδύνευσαν πάρα πολύ και πλήρωσαν με τη ζωή τους ε, γιατί πολέμησαν κατά της πολιτικής διαφθοράς. Ε, όλοι έχουμε καθήκον απέναντί τους. Αυτοί αγωνίστηκαν για την αλήθεια και για την ελευθερία. Αξίζει να αγωνιστείς μέχρι το τέλος. Ε, αλλά και εμείς ελεύθεροι δημοσιογράφοι και εσείς ε, θα πρέπει να υποστηρίξετε τα δικαιωμάτά τους. Ε, δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε ότι στην Ευρώπη πεθαίνουν δημοσιογράφοι για την αλήθεια. Δεν επιτρέπεται ούτε να ξεχάσουμε, ούτε να σιωπάσουμε. Δεν επιτρέπεται ούτε να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Χαίρομαι που ε, εγώ ε, μπορώ να κάνω αυτό το επάγγελμα για τους αναγνώστες μου ε, και δεν υποχώρησα μέχρι το τέλος απέναντι στον Τάγκνα. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Τοπολάγκα. Και ε, τώρα θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας παρακαλώ να μιλήσετε μόνο για τέσσερα λεπτά. Ο κύριος Άντριος Πυρκάουσκας. Thank you, Chair. Dear Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και αξιότιμα μέλη. Ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Ε, ακούσαμε πολλά προβλήματα από τις παρεμβάσεις των προλαλήσαντων. Να σας αναφέρω μερικά από τα πρακτικά μέσα και εργαλεία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει προβλέψει ένα κονδύλι για ε, ως πιλωτικό πρόγραμμα και προπαρασκευαστική δράση για την προστασία της ελευθεροτυπίας. Μπορεί να είναι μικρό το κονδύλι αυτό, αλλά πραγματικά είναι συμβολικό και μπορούμε να βοηθήσουμε καλά project για να ελαφρύνουμε λίγο ε, το βάρος που πέφτει στους ώμους των δημοσιογράφων. Ε, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, ε, κοιτούμε πώς ε, έχει η δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ακούσατε για το project ε, Πολυφωνία του Τύπου ε, που κάθε χρόνο ε, δημοσιεύει έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη και τονίζει και φωτίζει τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Και υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή και η νέα έκθεση καλύπτει τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα που αναφύονται και στο ψηφιακό κόσμο. Στη συνέχεια, δεν έχουμε μόνο διαρθρωτικά ζητήματα που καταδεικνύουμε, αλλά προσπαθούμε να βοηθούμε και μεμονωμένους δημοσιογράφους. Υπάρχουν διάφορα έργα που υποστηρίζουν ιδιαίτερα την ερευνητική δημοσιογραφία, βοηθώντας διασυνοριακά διασυνοριακές έρευνες δηλαδή δημοσιογραφικές και δημιουργώντας μέχρι και ξενώνες καταφύγια για τους δημοσιογράφους. Σήμερα απειλούνται και δικαστικά οι δημοσιογράφοι, οπότε παρέχουμε και νομική συνδρομή ε, από τα προγράμματα αυτά. Περνάει γρήγορα ο χρόνος. Να σας πω για το μέλλον. Προσβλέπουμε πάρα πολύ στην έκβαση των διαπραγματεύσεων των οργανικών για τη δημιουργική Ευρώπη, το Creative Europe. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα τέτοιο πρόγραμμα από εκεί ε, προβλέπει ειδικό προϋπολογισμό για την ελευθεροτυπία, την πολυφωνία του τύπου και ε, για ε, την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού περί των τύπων των εισαγωγικών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτά τα προγράμματα ε, ε, σε πολιετή βάση, πιο γερή. Και όταν θα έχουμε αυτά αποτελέσματα στο μέλλον, θα ξέρουμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Έχουμε ένα πρώτο γύρο σχολείων, ερωτήσεων. Το πολύ δύο λεπτά έκαστος παρακαλώ. Η κυρία Μετσόλα. Παρακαλώ. Thank you, Chair, very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Υπό τη σκιά της δοφωνίας της, ε, της ε, της κυρίας Γκαλίσια και του Κούτσια στη Σλοβακία. Υπό τη σκιά αυτών των δοφωνιών συζητάμε και της Τζο Κόξ που δολοφονήθηκε στον Ηνωμένο Βασίλειο πολιτικής και του Πάλεφτα Ντάμουι στο Γκτάνσκ. Στην περίπτωση της Δάφνης ε, δεν έχει συλληφθεί ο ένοχος και τα θέματα που ερευνούσε τα προστατεύει η κυβέρνηση. Δεν είναι αφηρημένα θέματα, αυτό λέμε. Είναι πραγματικές συνέπειες, θανατηφόρες συνέπειες. Πρέπει να πολεμήσουμε το μίσος και την παραπληροφόρηση όπου τα αντιμετωπίζουμε. Και το πιο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους τα μέσα είναι εξαιρετικά σημαντικά όπως και ο ανεξάρτητος διοικητικός κλάδος. Έτσι να το θεωρητήσουμε. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι ακρογωνίως λίθος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Κάτι παραπάνω από θεμελιώδης δικαίωμα είναι θεμελιώδης κανόνας ε, διακυβέρνησής μας. Αφορά το κράτο δικαίου. Το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο αυξάνεται και είναι πολύ ανησυχητικό είναι κάτι καλό να έχουμε ειδήσει στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορούν αυτά τα εργαλεία ε, να αποτελούν δικείμενο κατάχρησης. Και η κατάχρηση των metadata και των trolling και όλα αυτά επηρεάζουν την οτροπία του κόσμου και πουλάνε προπαγάνδα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα μέσα να καταπολεμήσουν το φαινόμενο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε φυσική προστασία δημοσιογράφων. Αναφέρθηκε αυτό αλλά επίσης και το, το, τις διάφορες μηνύσεις που αντιμετωπίζουν και θα πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά. Στην περίπτωση της Δάφνης, πολλές μηνύσεις έχουν κληρονομηθεί από τους γιους της. Και είναι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από πολιτικούς συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Ερώτηση. Αυτή η νομοθεσία κατά του ΣΛΑΠ, του Ευρωπαϊκού Νόμου, Πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για τους δημοσιογράφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε διάφορα εργαλεία. Μπορεί να μας ενημερώσει πού βρίσκεται όσον αφορά την νομοθεσία για αυτό το θέμα. Ζητήσαμε να μας πει η απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα έκανε. Καλή θα ήταν μια ενημέρωση για να προετοιμαστούμε και για την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Ζίπελ, να έχετε το λόγο. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω γερμανικά. Πιστεύω ότι δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι η δολοφονία ερευνητικών δημοσιογράφων και μετά από όσα ακούσαμε σήμερα δεν είναι παρά η οδυνορή ε, κορυφή του παγόβουνου που δείχνει την καταπίεση και την καταστολή των δημοσιογράφων. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να δούμε ε, ποιος υποφελείται από αυτά και ποιος ε, είναι ο ηθικός αυτούργος αυτών των δολοφονιών για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Το σημερινό πάνελ ξεκαθάρισε πόσο πολύπλευρες είναι οι πιέσεις και πόσο πολλές δυνατότητες έχει κανείς να απειλεί, να εκφοβίζει δημοσιογράφους και με πολύ ε, συγκεκριμένα μέτρα και οικονομικά να τους δυσκολεύουν τη ζωή και τη δουλειά τους. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο ε, οι δολοφονίες δημοσιογράφων, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε όταν αρχίζει αυτό το φαινόμενο να εκδηλώνεται, πώς θα προστατεύσουμε ε, τους ερευνητές δημοσιογράφους για να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο και χωρίς εμπόδια. Ερωτώ λοιπόν, Αυτό πώς θα το πετύχουμε. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία για τον τύπο. Χρειάζεται πιο αυστηρή νομοθεσία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την άσκηση επιρροής από πολιτικούς ή από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Χρειαζόμαστε άρα για πιο αυστηρούς κανόνες κατά της διαφθοράς και της άσκησης επιρροής. Ή μήπως από εκεί και πέρα χρειάζεται ευρύτερη πολιτική συζήτηση και με τους πολίτες για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και πόσο σημαντικά είναι τα ανεξάρτητα μίντια γιατί η ελευθεροτυπία και αξιόπιστες ε, πληροφορίες και ενημέρωση είναι πραγματικά εκ των όνων ουκάνευ για την ίδια τη δημοκρατία μας αλλά και για την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Και θα με ενδιαφέρει η άποψη όλων των ομιλητών νόμους. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε ή μήπως περισσότερο ε, συζήτηση για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, να αφυπνιστούν και να καταλάβουν τη σημασία του τύπου και να ε, συμπαρασταθούν ε, και να συμπαραταχθούν με αυτούς τους δημοσιογράφους που σήμερα απειλούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιόντσεβα. Merci pour me donner la parole. Euh, Ευχαριστώ τον Πατρίκ και την Τζούλη Μαζορτζάκ είναι οι ερωτήσει μου. Γενική γραμματέα, ο γενικό Γραμματέα του Κριστιαν Ζελουάρ, των δημοσιογράφων εγώ σύνορα, είπε ότι η... έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στη Βουλγαρία. Πάρα πολύ. Στη τελευταία έκθεση η Βουλγαρία είναι στην 110η θέση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Από το 2006 είμαστε στην... στο πολύ κάτω στη βαθμολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από εμά είναι χώρες οι οποίε δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βούλγαροι δημοσιογράφοι είναι στόχο του οργανωμένου εγκλήματος και των αρχών. Ο λόγο των επιθέσεων κατά των δημοσιογράφων είναι οι ερευνέ τους για τη διαφθορά, για τη συσχετισμό μεταξύ των πολιτικών και τη μαφία, για την καταχρηστική χρήση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που είναι γενναίοι διώχνονται από τη δουλειά του χάνουν τη δουλειά του υπό οποιοδήποτε πρόσχημα και δεν βρίσκουν πλέον δουλειά στην ειδικότητά τους. Υπάρχουν πολλά ονόματα όπως αυτά. Κάποιοι από αυτούς συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, όπως στο Γιάννοφ. Συνεχίζει η κυβέρνηση να διανέμει στα μέσα ενημέρωσης πώς τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως χωρίς διαφάνεια. Έτσι εγγυάται ένα περιβάλλον ε, που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν αρκεί η Ευρώπη να εντοπίσει την επιδείνωση της κατάστασης στη Βουλγαρία. Έχουμε την εντύπωση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα άφησαν τους δημοσιογράφους να πολεμούν μόνοι τους κατά της μαφίας. Αυτή η εντύπωση επικρατεί στη χώρα μου. Πώς εξηγείτε αυτή την πτώση της ελευθερίας του τύπου στη Βουλγαρία. Κατά πόσο είναι ανησυχητική η κατάσταση στη Βουλγαρία κατά την απόψή σας. Ποιο είναι υπεύθυνο κατά την άποψή σα για την επονίδιστη αυτή κατάσταση αφορά τα ΜΜΕ σε μια χώρα που είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σας ευχαριστώ. Ε, στη συνέχεια, Ρουίς Δεβέσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας. Γιατί πιστεύω ότι μας έδωσα μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα της ε, κατάστασης σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία. Θα ήθελα να αρχίσω ως εξής. Πιστεύω ότι η ελευθεροτυπία είναι κάπου το καύσιμο της δημοκρατίας. Τι εννοώ. Αν δεν υπάρχει αυτό το καύσιμο στη δημοκρατία ή αν δεν είναι το σωστό καύσιμο, η δημοκρατία μπλοκάρει. Γιατί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η ελεύθερη δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ενημέρωση. Γιατί η ενημέρωση μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη δημοκρατική άσκηση που είναι η διαμόρφωση άποψης ε, για να ε, αποφασίζουμε. Η δημοκρατία δεν είναι να ψηφίζεις κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά να ε, ξέρεις τι γίνεται. Και αυτό γίνεται με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ελεύθερα. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε από πολλές πλευρές αυτό το θέμα της ελευθερίας της ενημέρωσης. Όπως ακούσαμε σε μία από τις παρουσιάσεις, υπάρχουν δημόσια ΜΜΕ που στηρίζουν κυβερνήσεις και ιδιωτικά και χειραγωγούν φωτογραφίες. Άλλοι αναφέρθηκαν στην παραπληροφόρηση. Επίσης, ταυτόχρονα θα πρέπει να εγγυηθούμε πολυφωνία, πλουραλισμό στα μίντια και στα ιδιωτικά να υπάρχει διαφορετική ας πούμε συντακτική γραμμή και, να ε, εγγυηθούμε όχι μόνο ελευθεροτυπία για τα μέσα, αλλά και ελευθερία της έκφρασης γενικότερα. Και εδώ ε, συμπεριλαμβάνω και την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που και αυτή βάλεται και απειλείται. Η ακαδημαϊκή ελευθερία. Είδαμε στην Ιταλία πώς τιμώρησαν ε, μία ε, καθηγήτρια ε, που είχε στήσει ένα debate με φοιτητές και επέκριναν τον Σαλβίνη, την κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε πολύ πλευρά. Από τη μια έχουμε την καταπολέμηση της ε, παραπληροφόρησης και από την άλλη την προστασία των ελεύθερων και ανεξαρτήτων ΜΜΕ που είναι πραγματικά εκ των όνων κάνει για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια η κυρία Τοργίνο. Ταρντίνο. Η κυρία Ταρδίνο, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Μόλις ακούσαμε τη συνάδελφο που έλεγε ότι στην Ιταλία μια καθηγήτρια τιμωρήθηκε διότι οργάνωσε ε, ένα μάθημα στο οποίο αναφερόταν κατά του Σαλβίνη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα χειραγώγησης της πληροφορίας. Είμαι Ιταλίδα και επειδή είμαι από την περιοχή όπου αναφέρεται και συζητείται αυτό το θέμα, μπορώ να πω ότι αυτή η πληροφορία πραγματικά χειραγωγήθηκε. Αυτό το θέμα έχει σημασία, διότι σήμερα βλέπουμε με διάδοση των ψευδών ειδήσεων και είναι σημαντικό όχι μόνο οι δημοσιογράφοι να προστατεύονται απόλυτα, διότι είναι οι δικές μας πηγές, πρώτες πηγές πληροφοριών. Αλλά δεν πρέπει να χειραγωγούνται όμως οι ειδήσει απ' την άλλη από τα μέσα ενημέρωση. Ο τύπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπός κάλυψη γεγονότων και να έχει αφηγήματα που ίσως τελικά να είναι ψευδείς ειδήσει. Παραδείγματο χάρη σε αυτή την περίπτωση διευκρινίστηκε από την ίδια τη δασκάλα ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα θελημένο που προκλήθηκε από το Σαλβίνη. Θα πρέπει να στατεύσουμε λοιπόν τους, τις πληροφορίες, τους δημοσιογράφους και τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν δικαίωμα να έχουν σωστές πληροφορίε μέσω σοβαρών νομοθεσιών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό δεν μπορεί να υπαναχωρήσει, πρέπει να το κάνει. Ευχαριστώ. Επόμενος. Η κυρία Ντόνατ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε εδώ για να μιλήσετε για το σημαντικό θέμα. Έχω ερώτηση στα αγγλικά αρχικά και μετά ουγγρικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολλοί από εμά υποστηρίζουμε νομοθεσία κατά των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Πολλοί από εμά συμφωνούμε ότι πρέπει οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι να στηριχθούν. Οι φυσικέ απειλέ όμω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώ αντιμετωπίζονται, κανονισμό πλαίσιο για ποινικοποίηση απειλών κατά δημοσιογράφων θα βοηθούσε. Και να μιλήσω τώρα ουγγρικά, διότι η ερώτησή μου θα αφορά τον κύριο Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και αυτό που προσπαθήσατε να πείτε σε 10 λεπτά, να συνοψίσετε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουγγαρία. Όλοι έχουν δει τι γίνεται. Προσπαθούν να εκφοβήσουν τους δημοσιογράφους και να ε, αποφύγουν μια πραγματικά σωστή δημοσιογραφική και ερευνητική δουλειά. Αλλά δεν είπατε για τις ε, σωματικές απειλές και φυσικές που δέχονται οι δημοσιογράφοι, για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται, συχνά στην Ουγγαρία οι δημοσιογράφοι ε, ε, δεν μπορούν να εμπιστευτούν ούτε την αστυνομία. Δεν μπορούν να περιμένουν καμία βοήθεια από την αστυνομία έχετε στις υπόψεις σας καταγγελίες για τέτοια φαινόμενα. Καταγράφονται αυτά στην Ουγγαρία και τι μπορεί κανείς να κάνει για να τα αντιμετωπίσει. Thank you. The next one Ευχαριστώ. Η κυρία Φωνβίζε. Um... Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που υπόθηκαν από την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Έρχονται εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και ελπίζουμε ότι μετά θα υπάρξει άλλο ένα δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνω συγκρίσεις, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Την κατάστασή μας σε σχέση με τις δικές σας χώρες, όπως ξέρετε, είχαμε σημαντικό βαθμό παραπληροφόρηση χειραγώγηση των ψηφοφόρων και παρέμβαση από το εξωτερικό στο δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Εγώ δεν θέλω να διατείνομαι ότι η κυβέρνησή μου θέλει να παραπληροφορήσει τον κόσμο στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ανησυχώ όμω από το βαθμό παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων fakes, που υπάρχουν στα κοινωνικά μέσα που επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση στον Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα. Εσείς τι λέτε. Ποια είναι η εμπειρία σας. Ποιο είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο που λάβατε για να μειώσετε αυτού του είδους την παρέμβαση και την παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές σήμερα. Είναι μία από αυτές τις μέρες ε, που η ημερησία δεξί μας ε, συμπίπτει με την ε, πολιτική επικαιρότητα σήμερα ε, η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, θα μπορεί να κλείνει διάφορες ιστοσελίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης για λόγους δημόσιας τάξης με ένα διάταγμα αυτό προκειμένου να στραφεί κατά των πολιτικών αντιφρονούντων και να δράσει στο διαδίκτυο. Εμείς ε, σκεφτόμαστε ότι αυτό το διάταγμα που καθίσταται νόμος βάζει την Ισπανική κυβέρνηση εκτός ε, του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου του Μαΐου του 2018 για τον πλουραλισμό στα ΜΜΕ και την ελευθεροτυπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το ψήφισμα ζητείται από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν να απόσχουν από το να εθετήσουν μία απαραίτητα μέτρα που να περιορίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, στον μπλοκάρισμα mm. περιεχομένου και να μην, ε, υπάρχουν, να μην υπάρχει αυτόματη χρήση φίλτρων. Θέλουμε λοιπόν, λοιπόν, ε, κύριε Πένιξ, να σας ρωτήσουμε αν πιστεύετε ότι αυτό το, αυτός ο νόμος συνάδει με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και με τη Σύμβαση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για την κυρία Μάζερτσακ αναφέρατε μια σειρά δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν ή φυλακίστηκαν στα κράτη-μέλη. Όμως ε, δεν αναφερθήκατε στα τρία κράτη της Βαλτικής. Και θέλω να προσθέσω στον κατάλογο τρία ονόματα δημοσιογράφων στη χώρα μου που φυλακίστηκαν ε, για κάποιο καιρό, ε, είχαν περιορισμό, ε, Γιούρι Αλεξέιεφ, Βλαντεμίρ Λίτερπαν και Αλεξάνδρ Καπόνευκα. Επίσης, στην γειτονική χώρα στη Λιθουανία, για πάνω από ένα χρόνο βρίσκεται στη φυλακή ένας γνωστός δημοσιογράφος, ερευνητής δημοσιογράφος, Αργέτας Παλέτσκης ονομάζεται επειδή ερεύνησε τα γεγονότα του Ιανουαρίου του 1991. Ήδη του είχε επιβληθεί πρόστιμο για τα πορίσματά του, αλλά τώρα συνελήφθη. Και στις δύο χώρες κατέστη αυτό δυνατό λόγω τροποποίησης του ποινικού κώδικα. Δηλαδή ποινικοποιήθηκαν ε, πράξεις κατά των κρατικών συμφερόντων. Και αυτή η ευρεία διατύπωση, τα κρατικά συμφέροντα δηλαδή, μας ε, επιτρέπει να το οποιοδήποτε ερευνητής δημοσιογράφος και η... όταν ερευνά πράξεις των κυβερνώντων. Θέλω να θέσω λοιπόν μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν τώρα τέτοιες ε, τροποποίησεις του ποινικού κώδικα να εγκρίνονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρβανίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι είμαι δημοσιογράφος και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τους συναδέλφους μου, ευρωβουλευτή σήμερα, αλλά ο δημοσιογράφος είναι πάντα δημοσιογράφος. Θέλω να σας πω ότι η τελευταία μου περιπέτεια ήταν τα Paradise Papers, όπου οδήγησαν ουσιαστικά και στην απολυσή μου, όπως και άλλες απολύσεις που αφορούσαν ζητήματα καθημερινότητας. Για την Ελλάδα μιλώ. Βάζω ένα καινούργιο ζήτημα δεν έχουμε μόνο τα fake news. Έχουμε και τις αόρατες ειδήσει. Δηλαδή μεγάλα γεγονότα τα οποία κανείς δεν μπορεί να περάσει, να περιγράψει. Στην Ελλάδα σήμερα είχαμε αλλαγή, καθαίρεση μάλλον της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της κυρίας Στάνου, με μια χλιαρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό που έγινε και παραλλήλως έχουμε τέσσερις ιδιοκτήτες, ο οποίος ο ένας έχει εφημερίδες, εφημερίδες, όχι εφημερίδα, εφημερίδες, το πρακτορείο που τους διακινεί, δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, ένα συνδρομητικό κανάλι, μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, μία ποδοσφαιρική ομάδα και σχέση και με το στοίχημα. Έχουμε άλλους τρεις ιδιοκτήτες στην Ελλάδα. Όλοι έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες, όλοι έχουν άμεση σχέση με αυτό που λέμε εξουσία πού θα εργαστεί ο δημοσιογράφος. Πού θα μπορέσει ο δημοσιογράφος να κάνει όχι ερευνητική δημοσιογραφία που είναι σκληρή ιστορία, αλλά το αυτονόητο της κλασικής δημοσιογραφίας. Στην Ελλάδα ο Τεντέν σήμερα θα ήταν άνεργος. Δεν σας λέω για κάποιον επαναστάτη δημοσιογράφο, ακτιβιστή, για τον Τεντέν μιλώ. Βάζω λοιπόν ένα ζήτημα να το ξαναδούμε καθώς τα ανεξάρτητα δίκτυα, τα μικρά που υπάρχουν στην Ελλάδα, ή το Press Project που, ήταν, που είναι, ή το Left, ή ε, μικρά ή με, μεσαία site, δεν μπορούν να αντέξουν λόγω διαφήμισης. Τα πνίγουν. Μήπως λοιπόν το διοκτησιακό ζήτημα καθεστώς είναι ένα θέμα που πρέπει να επηρεάσει, να απασχολήσει, συγγνώμη, την Επιτροπή μας και ιδιαίτερα τη ΛΥΜΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ. Η κυρία Κάνκο, για δύο λεπτά. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους ε, για τις έντονες παρεμβάσεις σας. Μήπως ε, έγινε παρεξήγηση. Συγγνώμη. Should I... Νομίζω ότι είπατε Κούνκε. Μήπω έχετε οικογένεια στην Πορκίνα Φάσο που γεννήθηκα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είμαι συγκινημένη που περιβρίσκομαι σε αυτή την ε, ακρόαση για τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, και που ακούω τις ε, μαρτυρίες και τις παρουσιάσεις ιδιαίτερα από τους ανταποκριτές χωρίς σύνορα. Εμείς ε, είχαμε διάφορα προβλήματα στην Πουρκίνα Φασό με την ελευθεροτυπία και η πρώτη μου αντιπαράθεση με τη δημοκρατία ήταν ε, όταν ε, δολοφονήθηκε ο Μέτοράς μου και κάτι στην Πουρκίνα Φάσο το 1998 και τότε αρχίσαμε να πιστεύουμε στην ελευθερία του τύπου για τη δημοκρατία. Αν δεν είχε έρθει το RSF, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Έτσι λοιπόν, χάρη στο ΡΕΣΕΦ ε, τότε, ε, ήρθαν κάποιοι από το ΡΕΣΕΦ στην Μπουργκίνα Φάσο και ζήτησαν από την κυβέρνηση να ξεθάψει ε, το τόμα και να ξεκινήσει έρευνα. Γιατί αρχικά είπαν ότι ήταν ατύχημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα και κάποιο να καεί στο αυτοκίνητό του. Όταν ε, κάθεται εκεί δεν εξεράγει το αυτοκίνητο ότι υπήρχε άλλο αυτοκίνητο γύρω-γύρω. Πίεσε λοιπόν ε, η οργάνωση των ανταποκριτών χωρί σύνορα και εμεί μπορέσαμε ω φοιτητικό κίνημα να βασιστούμε σε αυτή την ε, υποστήριξη και χαίρομαι που σας τα λέω εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας πω την εξαιρετική δουλειά σας δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα και βοηθά τους ανθρώπους να μάθουν για τη δημοκρατία και μιλώ για γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν 20 χρόνια. Τότε δεν είχαμε όλη την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Για μένα η ελευθεροτυπία και η κυριαρχία των ΜΜΕ δεν ε, έχει σύνορα, ιδίω όταν ε, μιλάτε, παραδείγματο χάρη, για υποκλοπέ στα τηλέφωνα των δημοσιογράφων, ε, για κατασκοπία. Θα θυμάστε τι έγινε και στον Μαρκασούρη. αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση των δημοσιογράφων και οικονομικά στην Ευρώπη. Ε, και πολλές φορές τους λένε τι να κάνουν ε, και έχω και μία ε, κάπως προκλητική ερώτηση για σας. Είχαμε άρθρο στις εφημερίδες κατάπτωση του δημοσιογράφου λεγόταν. Έτσι λοιπόν, ε, πώς εξηγείτε τις δράσεις σας για να σώσετε τη δημοσιογραφία, γιατί υπάρχει και μια συνιστόσα ευθύνη ε, για την ποιότητα της δημοσιογραφικής δουλειάς. Thank you. And now... Σας ευχαριστώ, κύριε Φόξ. Sorry. Apologies. Μεγάλη μου χαρά να ακούω τις παρουσιάσεις για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Κατανοώ βέβαια όταν λένε οι άνθρωποι υπάρχει ανησυχία στην Ευρώπη για μια ρητορική κατατορμή μία ε, ε και ε, στρέφονται ο λαό ε, κατά τον mainstream ΜΜΕ. Νομίζω ότι είναι αλήθεια γιατί πολλοί πολίτες ε, αισθάνονται ότι δεν ε, τους υπηρετούν πλέον τα ΜΜΕ και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Και εγώ είμαι δημοσιογράφος και πριν γίνω ευρωβουλευτής ήμουν τμήμα τη φούσκα των ΜΜΕ και υπάρχει τέτοια φούσκα, πολλοί δημοσιογράφοι σκέφτονται το ίδιο. Είναι κάτι σαν ομαδικό και αν δείτε τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί δημοσιογράφοι δεν ε, ανέμεναν το κοινό της Βρετανία να ψηφίσει υπέρ του Brexit ε, και ε, δεν περίμενα ούτε τα μέσα στην Αμερική να ψηφίσουν όλοι ε, για τον, κάποιοι για τον Τραμπ και θα το ήξεραν αν έκαναν έρευνα και δεν ήταν μέσα στη φούσκα. Έτσι λοιπόν μπορεί να ε, τυφλωθούν από τον λαϊκισμό ε, τα μίντια. Και νομίζω ότι μερικές φορές η ίδια η δημοσιογραφία δεν είναι αρκετά ερευνητική αυτή τη στιγμή και ανησυχείται πάρα πολύ με τις απόψεις ε, μιας μικρής ομάδας ανθρώπων. Επίσης πιστεύω ότι ενίοτε είναι καλό να μετακινούνται από τα μαζικά ΜΜΕ οι άνθρωποι και να ε, στρέφονται σε εναλλακτικά ΜΜΕ. Τα ακούσαμε τι συνέβη στην Ουγγαρία. Μερικές φορέ πρέπει να δημιουργήσει κανεί εναλλακτικά μέσα ενημέρωση ε, για να πει την αλήθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριο τρόπος που ξέρουμε για τα κίτρινα γυναίκα στη Γαλλία δεν είναι γιατί το βλέπουμε στι ειδήσει στο BBC, αλλά γιατί έχουμε κάποιου πολίτε δημοσιογράφου που μα δείχνουν του Γάλλου δημοσιογράφου να ξυλοκοπούν του Γάλλου πολίτε. Επίσης, ε, είμαι κάπως ε, αγχώδης ε, για τους fact-checkers, αυτούς που ελέγχουν τα γεγονότα. Ανησυχώ για το αν μπορεί να υπάρχει μια επίσημη αλήθεια. Πώς ξέρουμε ακριβώς ποιος θα αποφασίσει τι είναι ακριβές και τι είναι αλήθεια. Άκουσα και στη σημερινή συζήτηση κάποιος να περιγράφουν την πληροφόρηση και τις ψευδοειδήσεις και το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξηγούσε ότι γιατί δεν ψηφίζουν οι άνθρωποι όπως ήθελαν να ψηφίσουν ε, και πολλές φορές ε, έχουμε θέσεις που έχουν προκαθαριστεί για να απαγορεύουν ε, πράγματα και νομίζω ότι αυτό σημαίνει επίθεση στην ελευθεροτυπία. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι χρειαζόμαστε ελευθερία, όχι περισσότερους κανόνες και κανονισμούς. Περί αυτού πρόκειται, περί ελευθερίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πάτρικ θα συνεχίσω στα πολωνικά. Ευχαριστώ. Ακούγοντας αυτά που είπατε, έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά, ισχολίστω με σημαντικά θέματα και σε ευχαριστώ για τα προβλήματα που είπατε για τη Σλοβακία. Είπατε καταπολεμήσετε την παραπληροφόρηση των πολιτών και χρησιμοποιείται επιχειρήματα παραπληροφόρησης όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία. Για παράδειγμα, για τα προβλήματα αναφερθήκατε στο βιβλίο του κ. Πιόντακ, ενός δημοσιογράφου, έγραψε κάτι για έναν πολιτικό. Ο πολιτικός χρησιμοποίησε το δικαίωμά του να προστατεύσει το όνομά του στο δικαστήριο. Και εσείς το χρησιμοποιείτε αυτό σαν παράδειγμα απειλής κατά της ελευθεροτυπίας. Ένας άλλος δημοσιογράφος μήνυσε τον κύριο Πιόντεκ και λήφθη απόφαση. Ήταν αρνητική η απόφαση κατά του κυρίου Πιόντεκ. Αποφασίστηκε και χρησιμοποιούσε ψευδείς πληροφορίες. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το παράδειγμα σαν παράδειγμα προβλημάτων με την ελευθερία του τύπου στην Πολωνία. Το ίδιο και με το δεύτερο παράδειγμα την υπόθεση των δύο πύργων στην Πολωνία. Κατέληξε στο Διοικητικό Δικαστήριο στην ε, Πολωνία πρόσφατα, ελήφθη απόφαση και έκλεισε η υπόθεση. Ξέρετε πώς κατέληξε αυτή η υπόθεση ή χρησιμοποιείται ο ίδιος παραπληροφόρηση κατά των παρισταμένων στην Επιτροπή. Ξέρετε πώς κατέληξε η υπόθεση. Αυτό που χρειαζόμαστε και που είναι σημαντικό όταν καταπολεμούμε την παραπληροφόρηση δεν πρέπει οι ίδιοι να παραπληροφορούμε τους πολίτες μας. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να περιμένουμε ότι οι πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ είναι υψηλής ποιότητας. Ζητούμε μια επαγγελματική συζήτηση, διότι αυτά τα δύο θέματα, αυτές οι δύο υποθέσει είναι πασίγνωστες για μα. Δύο αποφάσει δικαστηρίων αφορούν. Και γιατί δεν αναφερθήκατε σε αυτές. Αυτά που είπατε ήταν ε, παραπληροφόρηση κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Αδάμοβιτς. Η κυρία Αντάμοβιτς. Η κυρία Αντάμοβιτς, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε πολύ καλά παραδείγματα. Δυστυχώς, στην Πολωνία έχουμε πρόβλημα. Με την ελευθεροτυπία και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα κατάχρησης εξουσίας από πλευράς καθεστώτος αυτοί οι δημοσιογράφοι διώκονται. Ακόμα και αν τέτοιες υποθέσεις εκδικάζονται στα δικαστήρια, αυτές οι υποθέσεις απορρίπτονται. Η υπόθεση των δύο πύργων δεν έληξε ακόμα, διότι δεν έχουμε τελεσίδικη απόφαση. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος αναφέρθηκε στα βήματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε η ελευθερία του λόγου να προστατεύεται στην Ένωση. Αλλά πρέπει να πω και εγώ ήθελα να γίνει αυτή η ακρόαση και ήθελα να συζητήσουμε να προβληματιστούμε, να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε, να προστατεύσουμε την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, αλλά ταυτόχρονα να μην πέσουμε σε παγίδες, σε παραπληροφόρηση. Να χρησιμοποιούμε εκφράσεις μίσους. Πρέπει να χαράξουμε μια, κάποιο όριο. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το θέμα των λόγων μίσους, μισαλλοδοξίας. Ο κύριος Τέρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Τέρης, να ευχαριστήσω αυτούς που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Είμαι πρώην κομμουνιστική χώρα εγώ και ζούσα στη ΣΥΠΑ για πάνω από 16 χρόνια και είχα την ευκαιρία να δω πώς τα μέσα έδρασαν και αντέδρασαν σε πρώην κομμουνιστική χώρα και πώς έδρασαν και αντέδρασαν στη ΣΥΠΑ. Τι έμασα, τι έμαθα. Όλοι συμφωνούν ότι είναι η τέταρτη εξουσία τα μέσα ενημέρωση. Ο ρόλο του τη δικαστική εξουσία εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία είναι να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματα και ελευθερίε των ατόμων. Και αυτό είναι ο ρόλο των μέσων ενημέρωση σε οποιαδήποτε κοινωνία. Έχουμε πρώην συναδέλφους εδώ που αναφέρθηκαν στην παραπληροφόρηση, κακή πληροφόρηση, τα μέσα καμιά φορά είναι τυφλά, τυφλώνονται από το λαϊκισμό, είπε κάποιος συνάδελφος. Αυτή είναι η κατάσταση στη Ρουμανία. Αν συμφωνούμε ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωση είναι να αναφέρουν τα γεγονότα και να διαφυλάσσουν και προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων, τι είδαμε στη Ρουμανία επί σειρά ετών δημοσιογράφοι και οι φορεί των μέσων ενημέρωση αντί να προστατεύονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα των τα ατομικά βρίσκουν δικαιολογίε για τις καταχρήσει του κράτους κατά των ατόμων. Πολλά άρθρα στο ρουμανικό τύπο υπάρχουν όπου οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να βρουν δικαιολογίε για παραβιάση πλευρά των αρχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων. Παραδείγματα. Όλοι μιλάνε για τη Ρουμανία. Όποτε αναδύεται το θέμα της Ρουμανίας, το θέμα της δικαιοσύνης υπονοείται και τίθεται. Το 2016, κάθε χρόνο μάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωβαρόμετρο αποκαλείται. Το 2016, από το 2015 στο 2016, η εμπιστοσύνη του κοινού στη Ρουμανία για τη δικαιοσύνη μειώθηκε κατά 15%. Μεγαλύτερη πτώση εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό θεσμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά όταν ο κόσμος είναι αντικείμενο κατάχρηση από το κάτω, όταν οι δικαστές, οι μίκιο, οι άλλοι θέτουν τα θέματα κατάχρηση εξουσίας, αμέσως λένε οι δημοσιογράφοι γιατί εσείς υποστηρίζετε τους διεφθαρμένους, τους, λένε να σιωπάσουν. Αντί να συζητούν το θέμα, το θέμα καλύπτεται και εξατομικεύεται. Ερώτηση λοιπόν. Έχουμε εκπρόσωπο τον δημοσιογράφο χωρίς σύνορα. Δύο λεπτά, δύο δευτερόλεπτα μάλλον. Στην τελευταία έκθεση για τη Ρουμανία, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα είπαν ότι μυστικοί πράκτορες της Ρουμανίας ήταν άνω δημοσιογράφους και του παρακολουθούσαν. Σχόλιο σα. Ένα δημοσιογράφο στη Ρουμανία έγραψε κάποια άρθρα και έλεγε ότι καμιά φορά ακόμα και κατά πολέμηση διαφθορά δέχονται παράπλευρε απώλειε μιλώντας για ανθρώπους των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται. Πόσους δέχεστε εσείς να είναι αντικείμενο παραβίασης α, των δικαιωμάτων τους, να πέφτουν θύματα παραβίασης δικαιωμάτων για να καταπολεμήσουν διαφθορά. Ευχαριστώ για το Renew. Κύριε Σπέκα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιμέκα. Για το θέμα των ερευνητών δημοσιογράφων σχόλιο. Είμαι από τη Σλοβακία. Ο Γιάνν Κούτσα δολοφονήθηκε. Εδώ και ένα μισή χρόνο. Τραγικό γεγονός. Αλλά υπάρχει και θετική όψη. Δηλαδή η εξυχνίαση του εγκλήματος πρόδευσε. Πρόδευσε, πρόδευσε συγγνώμη. Και αποκαλυφθήκαν ε, η ανάμειξη των δικαστών, η διαπλοκή αποκαλύφθηκε. Και χάρη στην πίεση του Ευρωκοινοβουλίου, όλοι στη χώρα μου κατανοούν ποιο ήταν το έργο του Γιάνν Κούτσακ και ότι ο θάνατός του και η δουλειά του άλλαξαν τη Σλοβακία για πάντα. Αυτό εν είδη ενθαρρύνσεως προς τον κύριο Ταπαλάγκα και τους άλλους συναδέλφους, συνεχίστε να κάνετε τη δουλειά σας. Είναι σημαντικό, απαραίτητο για τη δημοκρατία μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας υποστηρίζει. Η κυρία Χούνκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, λέει η κυρία Κούνκε. Κύριε Πένδιξ, ποια είναι η βασική πρωτοβουλία από την πλευρά μα, από το Ευρωκοινοβούλιο, από τους ευρωβουλευτέ, Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Κυρία Μάγιατσακ, ποια νομική πρωτοβουλία χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να καταπολεμηθεί η ατιμορρησία εκείνων που δολοφονούν δημοσιογράφους ή απειλούν δημοσιογράφους. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης ε, της γνώμης προφανώς είναι το κλειδί της δημοκρατίας. Είναι προσφυλή σε όλους αυτά ε, και σε όλους μας και πολύ σημαντικά. Αλλά θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η γνώμη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ιδεολογία που να επιβάλλεται και όλοι να τη δέχονται. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία χωρίς ταμπού στην ανταλλαγή έκφρασης και γνώμης. Στην περίπτωση της Μάλτας τώρα και της Σλοβακίας δολοφονήθηκαν δημοσιογράφοι και προφανώς υπάρχει σοβαρή απειλή ε, και επίθεση ε, στην ελευθεροτυπία. Είναι πολύ σημαντικό και το τονίζω. Ταυτόχρονα όμως θέλω να αντιδράσω σε όσα λέγονται εδώ για την Ουγγαρία από το πάνελ που τα βρήκα εξαιρετικά μονομερή, ε, χειριστικά, χειραγώγηση και πραγματικά τρομακτική χειραγώγηση της ε, πραγματικότητας. Ε, ποια είναι τα γεγονότα, πώς έχουν τα πράγματα. Στην Ουγγαρία έχουμε ελεύθερη δημόσια συζήτηση, ζωντανή, ζωηρή, δουλεύει σωστά, έχουμε τοπικές εκλογές, ακούγονται διαφορές απόψεις, γίνονται debate, ήταν ελεύθερη προεκλογική εκστρατεία και το έδειξε και το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα ότι στην Ουγγαρία τα λέμε πιο πολύ έξω από τα δόντια από ότι σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι, δεν έχουμε ταμπού. Αυτό που άλλαξε τα τελευταία χρόνια είναι ότι τώρα έχουμε ε, δυνατότητες, κανάλια, ε, πόρταλ που, ε, που είναι συντηρητικά και δεν υπήρχαν στο προηγούμενο καθεστώς. Και αυτό ενοχλεί πολλούς στην αριστερά σήμερα. Εξού και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ε, που κάνουν επειδή είναι εξοργισμένοι και μάλιστα και προκλητικά αντιδρούν. Ε, για να καταλάβετε, με μεγαλύτερες τηλεοράσεις, πόρταλ και περιοδικά και εφημερίδες επικρίνουν την κυβέρνηση και καλά κάνουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει μια πολιτική ομάδα να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και να κατέχει την αλήθεια. Συζήτηση να γίνεται, ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει ε, να έχει ο καθένα την ελευθερία να έχει την πολιτική του γνώμη. Αλλά δεν είναι, ο κολεκτιβισμός δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία. Ο κύριος Τσεχοντάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά πίστευτο το άκουσα απόψε. Δεν φανταζόμουν ότι μπορούν να γίνουν αυτά σε ευρωπαϊκά κράτη. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι πάντοτε η στάση. Βέβαια, δεν συμφωνώ πάντοτε με όλα όσα ακούστηκαν, όμως υπάρχει ένα πρόβλημα ε, με την ερευνητική δημοσιογραφία. Εγώ Είμαι γιατρός ε, και πολλές φορές είδα δημοσιογράφους να έρχονται σε κατεπήγοντα περιστατικά. Ε, νομίζω και δέχτηκαν επίθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μία νέα στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είμαστε συνεκτικοί. Πρέπει να δώσουμε οικονομική στήριξη καταρχήν Επίσης, ε, έχουμε καταθέσει στο Βουλή της Ρουμανίας ένα νομοσχέδιο έτσι ώστε ένα ποσοστό ε, να γυρνά στους ε, ερευνητές δημοσιογράφους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε μέρα όταν αποκαλύπτουν υποθέσεις διαφθοράς. Νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να εκπονήσετε ένα κώδικα δεντολογίας που να διασφαλίζει αυτή την υποστήριξη. Γιατί, παραδείγματο χάρη, ε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να έχουμε ε, δημοσιογράφους δημοσιογράφου. Ε, κάτι άλλο θα μπορούσε να είναι μια πρόβλεψη νομική για όσους δέχονται επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ε, παραδείγματο χάρη, ο δημοσιογράφος ε, κινδυνεύει ε, τη ζωή του. Μπορεί να έχουμε, παραδείγματο χάρη, εκτός από ένα δημοσιογράφο και έναν αστυνομικό που κινδυνεύει τη ζωή του και αυτός προστατεύεται. Ε, νομίζω ότι και η ζωή του δημοσιογράφου θα πρέπει να προστατεύεται. Δεν έχετε και άλλες προτάσεις. Εγώ είμαι ανοιχτό. Εδώ θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία. να μην ξεχνάτε ότι και μία ψευδή είδηση μπορεί να οδηγήσει ε, σε δολοφονία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, γιατί τέτοια πράγματα δεν ε, τα ακούμε και δεν το πιστεύουμε ότι συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, κυρία Στρουγιάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω, κυρία Στρουγκαρίου. Να πω ότι συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια του κυρίου Τέρχες όταν ε, μίλησε για χειραγώγηση και για το ρόλο ορισμένων ε, τραστ με μία ε. γιατί ένα από τα πιο σημαντικά τραστ μη είναι ουσιαστικά στα χέρια του κυρίου Βοικολέσκου, ο οποίος πρέπει να πληρώσει ακόμα 60 εκατομμύρια στο ρουμανικό κράτος και έχει καταδικαστεί. Ε, και πολύ συχνά ε, πηγαίνει και στην, ε, στην έδρα του σταθμού. Εδώ είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και εκπρόσωπο της Κομισιόν. Και θέλω να ρωτήσω το εξή. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους ερευνητέ δημοσιογράφους και ακούσαμε ιστορίες και υπάρχουν και πολλές ακόμα. Γιατί το 2018 ε, συνελήφθησαν ε, ένας Ρουμάνος και ένας Βούλγαρος δημοσιογράφος ενώ ερευνούσαν ε, πώς δαπανόταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν ισχυρότερο μηχανισμό για να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους τρίτων χωρών. Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός, αλλά δεν έχουμε ένα μηχανισμό που να προστατεύει τους δημοσιογράφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκπρόσωπε τη Επιτροπή και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Περαιτέρω δράσεις, τρει προτεραιότητε. Πείτε μας πώς θα συνεργαστείτε στο να αντιμετωπίσετε την κατάσταση αυτή. Επίσης, να λάβετε υπόψη τη συστάση των συναδέλφων μου. Ε, συνάδελφος από τους ανταποκριτές χωρίς σύνορα ε, ανέφερε ένα μηχανισμό ενός κουμπιού πανικού που μπορεί να πυροδοτηθεί αμέσως αν γίνει κάτι εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης και άκουσα και για την Δημιουργική Ευρώπη. Πολύ ωραία που έχουμε τη σχετική χρηματοδότηση, όμω για τα 61 εκατομμύρια ε, που ε, ε, εκταμιεύονται μόνο για αυτά τα προγράμματα, για τη δημοσιογραφία δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε περαιτέρω κονδύλια για να μην βρίσκονται υποπίεση οι δημοσιογράφοι για την χρηματοδότηση των project τους. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Τώρα να στραφούμε στους ομιλητές και πάλι. Ξεκινήσαμε νωρίς σήμερα το πρωί και σε κάθε σημείο της ημερησίας διάταξης υπερβήκαμε το χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, που θα βάλετε τα δυνατά σα να μην μακρυγορήσετε. Ξέρω ότι ακούσατε πάρα πολλέ ερωτήσει, δύσκολε κιόλα, αλλά προσπαθήστε παρακαλώ να συνοψίσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Να ξεκινήσουμε τώρα. Θα πρότεινα τρία λεπτά ο καθένας ε, να πάρει το λόγο, γιατί πρέπει να ε, ακούσουμε και ακόμα τρεις ανθρώπους, στους οποίους θα θέσουμε ερωτήσεις. Ξεκινήστε κύριε Πένιξ, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά, αλλά να ξεκινήσω με το εξής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προλαμβάνουμε την παρενόχληση των δημοσιογράφων. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ποιοτική δημοσιογραφία και να προστατεύσουμε τους δημοσιογράφους. Και επανέρχομαι σε μία από τις ερωτήσεις εδώ. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς. Γιατί τώρα οι δημοσιογράφοι δεν έχουν πίστη ε, στους θεσμούς, ε, ούτε καν στις ενώσεις των δημοσιογράφων για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ζωτικό ζήτημα. Θα πρέπει να μπορέσουμε επίσης να ασκούμε διώξεις στα κράτη μας. που υπάρχουν ε, καταχρήσεις εξουσίας, θα πρέπει να μπορέσουμε να ασκούμε διώξεις. Επίσης, ε, θα πρέπει να το δούμε αυτά όλα υπό το κλίμα που κυριαρχεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει όλο ε, το θέμα ε, της κατάργησης του πλουραλισμού των ΜΜΕ. Όλο είναι και περισσότερο κινούμαστε ε, στο να υπάρχει μικρότερη προσοχή προς τις δημόσιες προς δημόσια τηλεόραση. Θα πρέπει να προωθήσουμε επίσης την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, γιατί πολλά θέματα σχετίζονται με αυτά. Δηλαδή, μιλάμε για την προστασία και την πρόθεση τη δημοσιογραφία. Είναι ο πρώτο πυλώνα. Δεύτερον, η βελτίωση των συνθήκων εργασία των μηχογράφων και διασφάλιση ε, του πλουραλισμού. Και επίση, ε, να προωθήσουμε την ερευνητική δημοσιογραφία και τον αλφαβητισμό στα ΜΜΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένο ρόλο να παίξει, γιατί πολλοί από εσά πήρατε το λόγο και είπατε. ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίως ίσως σε κάποια μέλη δίνουν πρωτοφανή κονδύλια. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επίσης έχουν ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά την πιθανή διαφθορά που μπορεί να προέρχεται από αυτό. Και εδώ πολλοί από τους δημοσιογράφους για τους οποίους συζητάμε ε, δέχτηκαν επίθεση ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει λοιπόν ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ένα μηχανισμό συναγερμού, ένα κουμπί εκτεκτονάγκης, αν θέλετε, αλλά θα πρέπει ε, ουσιαστικά όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν πολύ σύντομος. Κυρία Μάζερσακ. Ευχαριστώ. Σε τρία λεπτά να προσπαθήσω το ταχύτερο να το συνοψίσω για το ΣΛΑΠ. Δεν έχω το χρόνο να τα αναπτύξω. Επισημάνω την επόμενη εβδομάδα 12 με, στις 12 του μηνός, στις 18 και 30 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μια εκδήλωση που διοργανώνεται, όπου πολλές οργανώσεις υπεράσπισης ελευθεροτυπίας θα είναι παρούσες για να συζητήσουμε ακριβώς ποια μέτρα θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς οι Ευρωβουλευτές μπορείτε να εφαρμόσετε για να αντιταχθείτε ακριβώς στην χειραγώγηση των δικαστικών υποθέσεων, των εκδικάσεων υποθέσεων Στο θέμα τη χρηματοδότηση εξαρτήτων μέσων ενημέρωση, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα, χρειάζονται χρήματα, περισσότερα χρήματα. Γιατί την καταπολέμηση τη ατιμορρησία είναι ένα πραγματικό πρόβλημα όταν υπάρχει έλλειψη πολιτική βούληση και όταν οι δημόσιε αρχέ ε, συνδέονται, τα συλληπιτήρια και οι ομιλίε δεν αρκούν. Χρειάζεται πολιτική πίεση μεγάλη επί των χωρών όπου οι δημοσιογράφοι απειλούνται ένα κομβίον συναγερμού θα ήταν χρησιμότατο. Αν μπορούσε να επιφορτισμένος με αυτό ένας επίτροπος και να μπορεί να συνδέεται με τις ε, αρχές. Θα είχαμε φαινόμενο μόχλευσης αν είχαμε αυτό. Ισχυρότατο. Να επενθυμίσω ότι οι δημοσιογράφοι χωρί σύνορα έκαναμε ε, 10 προτάσει. Μπορούμε να τι υπενθυμίσουμε κάποιε από αυτέ. Υπάρχουν όλε εδώ. Ελάτε να πάρετε ένα αντίτυπο. Ευχαριστώ. Οι δύο δημοσιογράφοι μας, ο κύριος Άλελη, για τις απειλές. Τους τελευταίους δέκα μήνες αυξήθηκαν τα απειλητικά μηνύματα. 6,5 χρόνια υπάρχουμε, αυξάνεται η βία των απειλών, πλησιάσαμε τις αρχές, προσπαθήσαμε νομικά να το αντιμετωπίσουμε και φαρμόσαμε, δώσαμε κάποια πρωτόκολλα στο προσωπικό μας. Τι συμβαίνει, τι μπορούν να κάνουν είναι κάτι καινούριο για μας. Δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία. Ευτυχώς, πιθανότατα. Λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες. Περί ανταγωνισμού, Φερρυπίν. Όταν πάνω από 400 φορείς είναι υπό ένα πλαίσιο και μία ιδιοκτησία, Ίσως να υπάρχει κάποια προσέγγιση, κάποιος κανόνας. Βοηθάει αυτό τον ανταγωνισμό. Βοηθάει τον πλουραλισμό των απόψεων. Είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο να εξεταστεί. Αυτό είναι κάτι που δεν κάνουν οι Ουγγρικές αρχές και εσείς λακωνικότατο. κύριε Ταπαλάγκα. Τελευταίος, ευχαριστώ, όσον αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ε, οι ερευνητές δημοσιογράφοι ξέρουν τι κάνουν, έχουν υπομειστεί τις ευθύνες τους, χρειάζονται βοήθεια νομική, χρήματα για νομική αρρωγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρίσιμο. Παραπληροφόρηση για το Brexit που αναφέρατε κάτι μια ερώτηση. Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι ανέφικτη Δεν πα σταματήσει τη βροχή ούτε τον άνεμο. Μπορεί όμω να αποκαλύπτει πάντα την αλήθεια. πολέμηση τη παραπληροφόρηση σημαίνει αποκάλυψη τη αλήθεια καθημερινά. Και μακριά από τη Ρωσία. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, μακριά από τη Ρωσία. Τώρα ρουμανικά να απαντήσω στον κύριο Τέρχεσου. To be more για να είμαι πιο σαφής. Είπατε κυρία Τέρχες ότι υπερασπίσαμε τις ε, καταχρήσεις είναι ψέμα. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ο τρόπος ε, με τον οποίο το δικό σας κόμμα προσπαθεί να παρουσιάσει τους κατεδικασθέντες πολιτικούς ως θύματα που δεν είναι. Αυτό που δεν είπατε εσείς ε, και υποστηρίξατε τον κύριο Ντράγνα στο παρελθόν, ε, ασκήσατε ε, κριτική στον κύριο Ντράγνα και στο κόμματα πριν να φτάσετε ε, στους καταλόγους για να γίνετε ευρωβουλευτής, αλλά όταν σας έβαλαν στους καταλόγους σταματήσατε. Αυτό που δεν είπατε σε αυτό το κοινό είναι ότι πριν να είστε πολιτικός ήσασταν ιερέας. Και ως ιερέας τελικά υποστηρίξατε έναν άνθρωπο που είχε καταδικαστεί για κλοπή ψήφος και όπως ξέρετε είναι αμάρτημα η κλοπή. Μπορώ να απαντήσω. Συγγνώμη, ξανανοίξατε, ναι, αλλά ήταν μια προσωπική απάντηση. Να νομίζω ότι δικαιούστε να δώσετε μια σύντομη απάντηση. Και εξακολουθώ να είμαι η δεν υπεράσπιζα πολιτικούς, υπεράσπιζα το δικαίωμα κάθε Ρουμάνου πολίτη που κατηγορήθηκε από οποιοδήποτε κρατικό όργανο να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του, ανεξάρτητα από το άτομο αυτό ήταν ένας απλός πολίτης ή πολιτικός. Και πρέπει να δηλώσω ότι πέρα από τους πολιτικούς είχαμε χιλιάδες ε, πολίτες που δεν είναι γνωστά τα ονόματά τους, τον οποίο είχε καταστροφή ζωή και κάποιοι πέθαναν ε, και μετά το θάνατό τους ε, τους αθώωσε η δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, ποιος θα ξαναφέρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους, αυτή είναι η ερώτησή μου. Καλώς και ήσασταν σύντομος κι εσείς. Δεν μπορούμε. Κλείσουμε δηλώνοντας απλώς ότι αυτό είναι το τέλος της συζήτηση Είναι ανοιχτή η συζήτηση. Θα παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Για τα επόμενα χρόνια σίγουρα. Είναι κάτι διακομματικό, διασυνοριακό. Επικρατεί ανησυχία παντού όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης, πώς να καταπολεμηθεί μισαλοδοξία στο διαδίκτυο, εκτός διαδικτύου, αυτή η μόλυνση, αν θέλετε, όχι μόνο όσον αφορά τι πολιτικέ διαδικασίε εκλογέ, αλλά όσον αφορά την καθημερινή ζωή. Σας αποχαιρετούμε, ευχαριστώντας σας για τις προσπάθειές σας και που υποστηρίζετε αυτές τις σημαντικότερες αξίες για το θεματολόγιο του Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εσείς τα μέλη του πάνελ τιμάτε το Κοινοβούλιο ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό, εκ καρδίας. Ορίστε. Ναι, ναι, ναι, να χειροκροτήσουμε. Τους το οφείλουμε, τους ευχαριστούμε. Και ανακοινώνω ότι θα συνεχιστεί η ακρόαση με δεύτερο γύρο, με ένα δεύτερο πάνελ. Αποχαιρετούμε τα τέσσερα αυτά μέλη του πάνελ και καλούμε τα επόμενα τέσσερα μέλη του πάνελ παρακαλούμε να έρθουν εδώ στο βήμα να λάβουν τις θέσεις τους. said there's still one hour and a half to go. Έχουμε άλλη μια μισή ώρα μέχρι να τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Do it right and smooth. Πάμε γρήγορα. We welcome. Καλωσορίζουμε τα τέσσερα νέα μέλη του πάνελ για τη δεύτερη ενότητα ε, της ακρόασης. Που ε, τώρα θα ασχοληθούμε πώς να καταπολεμήσουμε ε, τη ρητορική μίσους online και offline και την παραπληροφόρηση. Καλωσορίζουμε την κυρία Μάγια Μαζουρκίεβιτς που εκπροσωπεί το Alliance for Europe, ένα δίκτυο πολιτών. Καλωσορίζουμε τον κύριο Διέγο Ναράγχο ε, που εκπροσωπεί την European Digital Rights, τον Ντανιέλ Μίλο από το Globsec Policy Institute και την κυρία Κάτριν Χούγκεντούμπελ Διευθύντρια στο ILGA Europe. Αρχίζουμε λοιπόν. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις όσοι προλάβουν. Δίνουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Μαζουκίεβιτς, Alliance for Europe, για τα επόμενα 8 με 9 λεπτά, αν μπορείτε. Λιγότερο από 10. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μάγια Μαζορκίεβιτς, εκπροσωπώ την πλατφόρμα Alliance for Europe, η πλατφόρμα για συνεργασία φιλοδημοκρατικών και φιλοευρωπαϊκών οργανώσεων. Και είμαι και συντονίστρια του Keyword Warriors, ε, offline και online για καταπολέμηση των ε, fake news, της παραπληροφόρησης στη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μιλήσω για την παραπληροφόρηση και τη ρητορική του μίσους. Ε, έχουμε το, εξα... το παράδειγμα της Πολωνίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό συμβαίνει σχεδόν παντού, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα η Πολωνία εδώ. Τι θέλω να πω εδώ μιλάμε για το εδώ και τώρα, ε, ότι αυτά συμβαίνουν εδώ και τώρα, αλλά αφορούν το μέλλον μας. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, αν δεν καταλάβουμε ότι χρειάζονται τα χρήματα για να καταπολεμηθούν αυτά τα φαινόμενα παραπληροφόρησης, μπορεί και σε 10 χρόνια από τώρα ε, να χρειαστεί να ε, παλεύουμε πολύ σκληρά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στην Πολωνία 80-90% του λαού ε, ε, είναι υπέρ της Ευρώπης, αν τους ρωτήσετε. Είναι από τα πιο φιλοευρωπαϊκά έθνη η Πολωνία στην Ευρώπη. Shift of attitudes. Ε, είναι δυνατόν να αλλάξει η συμπεριφορά. Το 2015, στην αρχή του 2015, πριν όλες τις εκλογές προεδρικές και βουλευτικές, η Πολωνία ήταν υπέρ των ε, προσφύγων. Αλλά ξέσπασε μια προπαγάνδα στα μίντια και οφείλονται και πολιτικοί γιατί ήταν ιδιοκτήτες των μίντια. Άλλαξε η συμπεριφορά. Ήδη από το τέλος του 2015 βλέπετε ε, ε, ότι πάνω από τους μισούς Πολωνούς δεν ήθελαν πια να δεχθούν πρόσφυγες. Αυτό μπορεί να αλλάξει λοιπόν και στη στάση τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τέλη του 17 το Δεκέμβριο έγινε ε, μια έρευνα από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών. Στην ερώτηση τι θα κάνατε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σας ανάγκαζε να έρθουν πρόσφυγες στην Πολωνία, 51,2% είπαν ότι θα ήταν αντίθετοι, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε λοιπόν τα συναισθήματα πώς ε, να κινούνται κατά των προσφύγων και των μεταναστών. Η προπαγάνδα επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτονται οι Πολωνοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι βλέπουμε στο διαδίκτυο για τους ε, πρόσφυγες. Ήδη από το 2015 και πιο πριν. Φόβο, χειραγώγηση και παραπληροφόρηση. Και εδώ μπορούμε να δούμε διάφορα παραδείγματα του τι βρήκαμε στο διαδίκτυο, γιατί το παρακολουθούμε και κοιτάμε τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε εικόνες κατά των προσφύγων, κατά των μεταναστών που δουλεύουν με τα ε, συναισθήματα του κόσμου, με το θυμικό. Τα περισσότερα είναι και τα ψέματα και ε, στημένα. Πρόσφατα τι είδαμε και από το ο Κατσίνσκι, ο Γιάροσλαβ, ε, ο ηγέτης του κόμματος του ΠΙΣ, λέει ότι φαίνουν εξωτικά νοσήματα οι ε, πρόσφυγες και ότι εμείς ε, φοβούμαστε οτιδήποτε δεν ξέρουμε οι Πολωνοί. Το ίδιο έγινε και με τους πρόσφυγες. Οι τεχνικές και τα εργαλεία της προπαγάνδας βάζουν τους πρόσφυγες αντιμέτωπος. Και χτες έλεγαν ότι στο Μόναχο ξέσπασαν ε, ταραχές και επεισόδια ε, ε, με μετανάστες που τα, τα ανακοίνησαν μετανάστες. Αυτά ήταν τελείως fake. τα καταρρίψαμε ως keyboard warriors. άλλη πληροφορία που μπορείτε να βρείτε από το 2017 είναι για τις περιφέρειες της Σαρία λέει και τις απαγορευμένες ζώνες. Πολύ συχνά το βλέπουμε από το 17, το επαναλαμβάνουν και πολιτικοί και τα διάφορα μέσα ενημέρωσης και πολλοί συζητούν για το παράδειγμα της Σουηδίας και λένε ψεύδι ουσιαστικά για το τι συμβαίνει στην Σουηδία. Ότι έχουν εκεί, ξέρω εγώ, 13 βιασμούς την ημέρα σε περιοχές που έχει πολλούς πρόσφυγες. Τι μπορούμε να δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας είπαμε, παρακολουθούμε το διαδίκτυο. Εμείς και το Ίδρυμα Battery πριν από λίγες εβδομάδες άρχισαμε να κοιτούμε τι λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 87% ε, των σχολείων που γράφουν οι χρήστες του διαδικτύου είναι αρνητικά αν το εξετάσεις βαθύτερα, τα περισσότερα από όσα αναφέρονται είναι επίση ψευδή. Όπως σας είπα, η Πολωνία είναι από τις πιο φιλοευρωπαϊκές ε, χώρες η Πολωνία. Αλλά τώρα το 87% των σχολείων που γράφουν στο διαδίκτυο είναι αρνητικά για την Ένωση. Και ο κόσμος τώρα πια πληροφορείται από το διαδίκτυο. αν ρωτήσει κάτι στο ίντερνετ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σου έρθουν αρνητικά σχόλια ή ψευδή. Κάτι που επαναλαμβάνουν πολλοί οι Πολωνοί πολιτικοί, ότι πληρώνει η Πολωνία περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι η Ένωση στην Πολωνία. Αν το γκουγκλάρετε αυτό στην Πολωνία, ε, ε, θα σας βγάλει το Google στις περισσότερες περιπτώσεις ότι αυτό ισχύει. Αυτό είναι ψευδέστατο. Ε, τώρα θα ήθελα να σας δείξω τα πιο δημοφιλή θέματα που απασχολούν τους Πολωνούς. Ε, εκεί παρακολουθούμε το διαδίκτυο για την παραπληροφόρηση και πριν τις βουλευτικές εκλογές η έκθεσή μας θα βγει τέλη Νοεμβρίου. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν, ότι η περισσότερη παραπληροφόρηση αφορά ε, θέματα ΛΟΑΤΚΙ, αντισημιτισμό, τους ξένους γενικά όχι μόνο πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά κυρίως και η οικολογία. Δηλαδή θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή ε, και και ένα ατύχημα που έγινε ε, στο βιολογικό καθαρισμό στην ε, Βαρσοβία και κυριάρχησε στην προεκλογική καμπάνια. Στη Γερμανία επίσης παρακολουθούμε τι συμβαίνει, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι απασχολεί τον κόσμο, έτσι, μια συνολική επισκόπηση. Σε πολλές χώρες τα θέματα της παραπληροφόρησης είναι εφάμιλα. Στη Γερμανία επίσης ε, αφορά τους ξένους, την οικολογία, τους μετανάστες και την ελευθερία του λόγου. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι εκλογές, ο αντισημιτισμός, οι μετανάστες, ε, οι εκλογικές συμμαχίες και ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζει ο κόσμος, ένα δημοψήφισμα δηλαδή. Ένας συνάδελφος που εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι τα μόνα, οι μόνες ειδήσει που δεν είναι fake news ε, στα μέσα ε, της ε, Μεγάλης Βρετανίας είναι τα νέα για τον καιρό και για τα αθλητικά. Όλα τα άλλα είναι fake. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουμε πρόβλημα και μας λένε ότι η πηγή όλων των δεινών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ένα ουράνιο τόξο και μας στέλνει όλα τα δεινά και στην Πολωνία και αλλού. Ε, ο νέος εχθρός στην Πολωνία τώρα είναι η Ολάτκη. Έχει γίνει viral από το Φλεβάρι. Λοάτκι... Α. Ανακοινείται πολύ το θέμα αυτό στον τύπο και πραγματικά αναφέρεται στο θυμικό Υποτίθεται ότι τα σχόλια είναι ουδέτερα, αλλά αν το ψάξουμε, ε, διαπιστώνουμε ότι δεν καθόλου ουδέτερα, είναι πολύ αρνητικά. Ε, απλώς, αν ψάχνεις με αρνητικές λέξεις, ε, δεν στο βγάζει ότι είναι αρνητικό. Είναι τεράστια επίσης η κάλυψη και η απήχηση. Τον Ιούλιο, όπου ήταν στο αποκορύφαμα, θα σας δείξω τι έγινε τότε στην Πολωνία, περίπου 400.000 χίτ είχε επισκέψεις ε, ε, αυτή η ιστορία με τα σχόλια. Ε, εδώ βλέπουμε τις λέξεις κλειδιά. Τι λένε λοιπόν ε, για τους ανθρώπους που ανήκουν σε μειονότητες οι Πολωνοί. Ε, τους συνδέουν με παιδεραστία. Ε, λένε ότι σεξουαλικοποιούνται τα παιδιά από την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Και όλα αυτά που συμβαίνουν δεν συμβαίνουν μόνο στα social media αλλά και στα κοινωνικά. Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου ε, είχε ένα ρεπορτάζ τηλεόραση ε, για τους ΛΟΑΤΚΙ προπαραμονή των εκλογών και λίγες ώρες πριν ε, σταματήσει η προεκλογική εκστρατεία. Και ήταν και στις 8 το βράδυ που είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση γιατί στις 8.30 έπαιζε η Εθνική Πολωνία στο ποδόσφαιρο ισχυρίστηκαν ότι συνέβη κάτι στην Πολωνία, ενώ δεν συνέβη, ήταν σε άλλη χώρα και έλεγε ότι οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ πληρώνουν τους ανθρώπους για να εκδηλωθούν. Εδώ βλέπετε ένα φωτομοντάζ για ε, ε, ε, το δήμαρχο της Βαρσοβίας που είναι ομοφιλόφιλο και είναι γνωστό αυτό και του κάνανε ένα φωτομοντάζ στο Gay Pride το 22 με 29 Ιουλίου έγιναν επεισόδια και το ήξερε η αστυνομία ότι θα γίνουν. Είχαν προετοιμαστεί για τρομοκρατική επίθεση κιόλα. και έγινε μεγάλη καταστολή ε, στο Gay Pride. Ε, πραγματικά αυτή η ρητορική μίσους υπάρχει και επηρεάζει πολύ ε, σημαντικά και πολύ αρνητικά. Και όπως ακούσαμε προηγουμένως, δολοφονήθηκε ο δήμαρχος ε, στο ΚΤΑΝΣΚ, ο Πάβελ Αντάμοβιτς, ακριβώς λόγω ρητορικής μίσους. Αυτό το είπε ο Δήμος ε, του ΚΤΑΝΣΚ, ότι η κρατική τηλεόραση, το, το TVP, πέντε φορές τη μέρα, 1700 τόσες φορές καταφέρθηκε κατά του Οντάμοβιτς και τον σκοτώσανε. Σας ευχαριστούμε για τις ε, πλήρε παρουσιάσεις σας. Πολύ εντυπωσιακή παρουσίασή σας, ε, ιδιαίτερα ολοκληρωμένη. Αλλά θέλουμε να έχετε κατά νου ότι είστε τέσσερις. Και κατόπιν ε, πρέπει να έχουμε και τις ερωταπαντήσεις. Να προσπαθήσετε να μην μακρηγορείτε, παρακαλώ. Ο κύριος Διαγώνα Ράγχο έχει το λόγο που εκπροσωπεί το EDR, European Digital Rights. Είμαστε ένα δίκτυο 42 ΜΚΟ που υπερασπίζουν online τα ψηφιακά δικαιώματα. Αν είχαμε ένα μότο για τη ρητορική μίσους, θα λέγαμε μισούμε τη ρητορική μίσους και μας αρέσει η ε, ελεύθερο η ρητορική. Αλλά υπάρχουν και κάποιες αποχρώσεις. Καταρχήν, για το περιεχόμενο υπάρχει πολιτική όθηση να έχουμε περισσότερες ευθύνες ε, οι πλατφόρμες ε, για να αστυνομεύουμε ε, το περιεχόμενο online σε οριζόντιο επίπεδο. Έχουμε την μελλοντική πράξη DSA και έχουμε και την οδηγία για το copyright και το κανονισμό για τα πτυκοκοστικά μέσα και έχουμε και έναν κώδικα τον κώδικα πρακτικής για τη ρητορική μίση Είναι διάφορε που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Όμω ε, δεν φαίνεται αυτό να έχει πραγματική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, το feedback που λάβαμε ε, από τον κώδικα δεντολογία δεν μα έφερε στοιχεία αξιόλογα το παραδέχτηκε και η Κομισιόν. Μέσα στο νομικό πλαίσιο βλέπουμε ότι αναζητούν πληροφορίε ε, επίσημοι και ανεπίσημοι φορεί. Ε, θα δείτε ότι έχουμε επίσημους, ε, επίσημα μέσα τον Donald Trump, το Fox News, το Vox, το Ισπανικό Κόμμα που είπαν ότι οι πρόσφυγες μπορεί να βιάσουν ε, γυναίκες ε, τρεις φορές περισσότερο σε σχέση με άλλους πληθυσμούς. Και επίσης έχουμε και μη μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, εδώ έχουμε τα πιο δύσκολα προβλήματα με τη ρητορική μίσους. Η ρητορική μίσους είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του διαδικτύου. Οι πιο σύγχρονες μορφές ρητορικής μίσους είναι μηνύματα που ε, μπαίνουν στην mainstream, στην παραδοσιακή πολιτική ε, και τελικά θέλουν ε, να δημιουργήσουν μια ψευδέστηση νομιμότητας και υποστήριξης για τον αγώνα τους. Έχουμε ρατσισμό, ξενοφοβία, έλλειψη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία φαίνεται να είναι σε αύξηση σε δημοκρατικά κόμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε δύο κύρια προβλήματα. Το ένα σχετίζεται με τη δυσκολία του κράτου δικαίου να προσαρμοστεί στι νέε τεχνολογίε ε, και το δεύτερο με το επιχειρηματικό μοντέλο των ε, υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Σε σχέση με το πρόβλημα του κρατή δικαίου υπάρχει τεράστιο μέγεθο πληροφοριών. Κάθε 60 δευτερόλεπτα έχουμε 3 εκατομμύρια από στο Facebook, ε, μισό εκατομμύριο tweets και έχουμε και άλλο υλικό. Μιλάμε για τεράστιο τεράστιο αριθμό πληροφοριών και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωνευτούν. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν ε, χειρονακτικά ε, να ελέγξει κανείς το περιεχόμενο. Και τι συμβαίνει. Η πλειονότητα των αποφάσεων λαμβάνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Αυτές οι ιδιωτικές οντότητες βασίζουν ε, την ε, απόφασή τους ε, σύμφωνα με τους όρους που περιέρχονται στο συμβόλαιό τους και βλέπουμε τελικά ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί ένδικων μέσων, βλέπουμε αυθαίρετες, αυθαίρετα κατεβάσματα σελίδα και διάφορα πρότυπα που βασίζονται κυρίως στην Αμερικανική νομοθεσία και στον δεντολογικό κώδικα. Θα ήθελα να δω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, ακούσαμε ότι ε, η ρητορική μίσους αφορά κυρίως τις αριστερές ε, απόψεις. Ε, δηλαδή αυτοί που δεν υποτίθεται ότι πρέπει να διαδίδουν τέτοιες απόψεις. Έχουμε και μια ομάδα Women on Waves που μπλοκαρίστηκε στο YouTube 30 ε, μέρες πριν από το δημοψήφισμα ε, για την άμβλωση στην Ιρλανδία και αυτό μας δείχνει ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στις μειονότητες και στις γυναίκες, στους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά και σε άλλες παρόμοιες ομάδες. Αυτό το πρόβλημα διευρύνεται από την κύρια ε, προσέγγιση ε, για, την, ε, για τον έλεγχο του περιεχομένου. Χρησιμοποιούν αυτά τα φίλτρα που μπλοκάρουν ή διαγράφουν περιεχόμενο. Ο κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση τι σημαίνει ότι απλώς καταργείται ένας αριθμός λογαριασμών και post και δεν υπάρχει καμία δράση καμία έρευνα, με συγχωρείτε. Επίσης, ε, τα φίλτρα αυτά δεν μπορούν να κάνουν αυτού του διαχωρισμούς. Ε, υπάρχει, τόσο χάρη, περίπτωση να κατεβαίνει νόμιμος λόγος ε, με αυτές τις τεχνολογίες. Ένα άλλο πρόβλημα που είναι ακόμη πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε είναι η έλλειψη εναρμονισμένου ορισμού της ρητορικής μίσους. Μία από τις εκθέσεις που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μα έδειξε ότι έχουμε πολλέ αποκλήσει μεταξύ τη νομοθεσία στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρά τι προσπάθειε τη Ένωση να του εναρμονίσει. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο, ε, ουσιαστικά η βλάβη δεν προέρχεται από το ίδιο το περιεχόμενο τις περισσότερες φορές, εκτός και αν πρόκειται για υλικό παιδικής ε, πορνογραφίας, αλλά από το πόσο μακριά φτάνει αυτό το περιεχόμενο, σε πόσο απευθύνεται. Ε, πολλές εταιρείε ε, έχουν τεράστια κέρδη μέσω από την εμπορική επιτήρηση και αυτές ε, οι εταιρείε φοβούνται ότι ε, θα γεμίσουν τις τσέπες τους με τη δική σου προσοχή, δηλαδή όσο περισσότερα κλικ γίνονται σε μια πλατφόρμα. Ε, ο CEO του Netflix είπε ότι δεν ε, υπάρχει άλλη εταιρεία ε, που να καλύπτει την ανάγκη σου όταν πηγαίνεις στο κρεβάτι. Γι' αυτό σου ε, στέλνουν το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Εκτός αν το σταματήσεις. Στην περίπτωση του YouTube υποθεί ότι όσο πιο προκλητικό είναι το υλικό, τόσο μεγαλύτερη η προσοχή δίνεται και τόσο περισσότερο χρόνο ξοδεύει στην πλατφόρμα και τόσο μεγαλύτερα τα κέρδη της πλατφόρμας και για τους ε, αριστερούς ε, ε, όταν λέω αριστερούς αναφέρουμε στην άκρα αριστερά τι συμβαίνει αρχίζουν να ψάχνουν υλικό και της ακροδεξιάς Τώρα, το πρόβλημα αυτό το επιχειρηματικό είναι ότι αυτοί αποφασίζουν οπότε πώ σε οδηγούν, αλλά ένα και περισσότερο, σε υλικό πληροφόρηση και υλικό μίσου προκειμένου να παραμένει στην πλατφόρμα. Προκειμένου λοιπόν αυτοί να σου πουλήσουν διαφημίσει ή να αγοράσει ε, πράγματα που δεν χρειάζεσαι. Θα προτείνω κάποιε λύσει στην παρουσίασή μου. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη με παρουσίασε κάποιε πολύ συγκεκριμένε λύσει που θεώρησα πολύ θετικέ. Θα το αφήσω λοιπόν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά ένα από τα πράγματα που θέλω να προσθέσω είναι η πολιτική της προσέγγισης. Η προσέγγιση της πολιτικής επικεντρώνεται στα συμπτώματα του προβλήματος και όχι στην αιτία του προβλήματος. Η λύση δυστυχώς είναι πολύ πιο δύσκολη από το να έχουμε ένα άρθρο ε, που να λέει ότι θα αντιμετωπίσει ρητορική τριτορική στο facebook. Μην ανησυχείτε, η λύση στο πρόβλημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ε, ουσιαστικά τοποθέτηση κατά του μίσους και της μισοδελοδοξίας ε, και να τοποθετούμαστε κατά του λόγου της ακροδεξιάς όπως βλέπουμε και στην Ισπανία. Επίσης, ε, κατάρτιση για τους υπαλλήλους και τα δημόσια πρόσωπα και να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός των ΜΜΕ. Μερικές φορές όταν η ρητορική μίσους βέβαια θα πρέπει και να τιμωρείται. Παραδείγματο χάρη όταν ε, έχουμε παρακίνηση σε γενοκτονία. Ε, επίσης όταν υπερασπίζει κάποιος ε, λόγο που παρακινεί σε έχθρα ή σε άσκηση βίας. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ποιος είναι ο μιλητής, είναι καλλιτέχνη, είναι πολιτικός, ποιο είναι το πλαίσιο, ποιο είναι ο σκοπός, ποιο είναι το κατόπιν κατόφλι της ε, αυστηρότητας. Ε, δηλαδή μπορεί να οδηγήσει ο λόγος αυτό σε πραγματική διάκριση ή σε δράσεις ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας, γιατί οι άνθρωποι ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλες πλατφόρμες και όχι αυτές τις σύνηθες τα τελευταία μου λόγια θα πρέπει να, να στραφούν σε άλλους τρόπους να αποφύγουμε την περιπληροφόρηση. Ε, στην Ισπανία έχουμε εθνικές εκλογές, παρακαλώ να πάτε να ψηφίσετε. Θέλουμε να αφήσουμε την ακροδεξιά σε μια σκοτεινή γωνία της ιστορίας, εκεί όπου ανήκει. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Ναράγχο. Σας ευχαριστούμε όλους ιδιαίτερος. Ο κύριος τώρα, Ντανιέλ Μίλο. Μάιλο Μίλο, πώς σας. Ντάνιελ Μίλο. Από το Globsec Policy Institute. Για ένα δεκάλεπτο το πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είμαι ερευνητή στο Globsec Policy Institute, κέντρο προβληματισμού στην Ευρώπη. Ασχολούμαι με θέματα εξωτερική πολιτική ασφαλεία, αλλά εξετάζουμε και τον αντίκτυπο που έχει παραπληροφόρηση και η παροχή πληροφοριών στη δημοκρατία και στις κοινωνίε μα εν Η Σλοβακία βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, είναι γείτονα της Ουκρανίας και λόγω γραφική εγκύτητα βλέπουμε εντοπίσαμε την παραπληροφόρηση και τα fake news πριν χτυπήσουν την Δυτική Ευρώπη και τι άλλε χώρε. Από αρχές του 2014, στην ακμή των μαχών στην Ουκρανία, διάφορε παραπληροφορήσει δόθηκαν και διάφορε πηγέ συνωμοτικέ εμφανίστηκαν στη Σλοβακία και σε άλλε χώρε περιοχή από το διαδίκτυο, διαδιόφωνο στο διαδίκτυο μέχρι περιοδικά πολυτελεία, κίτρινο τύπο, διάφορα μέσα ενημέρωση, διέδιδαν ψευδεί πληροφορίε. Ευτυχώ, στη Σλοβακία μάθαμε το μάθημά μα όσον αφορά το αυταρχικό καθεστώ του τότε Πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Μετσιάρ τη δεκαετία του 90 που σχεδόν κατάφερε να σταματήσει την ένταξη της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα έπεσαν κρίσιμο ρόλο στην πάλη για τη δημοκρατία. Και είμαι περήφανο να εκπροσωπώ εδώ το GLOBSEC που είναι ένα οργανισμό ο οποίο έγινε ένα από τα ηγετικά κέντρα τεχνογνωσία όσον αφορά την παραπληροφόρηση και τρόπου τρόπους αυτή στην Ευρώπη. Για να δείξω πού βρισκόμαστε τώρα και τι δυνάμει πρέπει να αντιμετωπίσουμε, α ξεκινήσω με μια παράθεση. Υπάρχει ένας Εβραίος πίσω από τα πάντα. Δεν θέλω να προσβάλλω αυτή την εθνοτική ομάδα. Είναι πολύ επιδέξη, έξυπνη, φιλόδοξη, κυρίως όσον αφορά αυτούς και τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Και πάντα είναι τεράστια, εκατομμύρια δολάρια είπα, έλεγχος χωρών. Γιατί να πολεμήσει κανείς όταν μπορεί να πετύχει τον ίδιο στόχο με άλλα μέσα, με τη χειραγώγηση ανθρώπων. Πιστεύετε ότι αυτή η παράθεση είναι από το Mein Kampf ή κάποιο άλλο φυλάδιο αντισημητικό ιστορικής αξίας. Όχι. Είναι από τον Ιανουάριο του 2019 από τη Σλοβακία. Και συνεχίζει και λέει γίνονται προεδρικές εκλογές ευρωπαϊκέ εκλογέ και του χρόνου εκλογέ για το Εθνικό Κοινοβούλιο τη Σλοβακία. Α προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε κάποιε βασικέ πληροφορίε και γεγονότα ότι εκείνοι δηλαδή, οι Εβραίοι, έχουν τεράστια δύναμη, διότι εκείνοι προφανώ ελέγχουν τα βασικά μέσα ενημέρωση και αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο και το λαό. Οπότε να ψηφίσουν υποψήφιους που κανονικά δεν θα μπορούσαν να πετύχουν σε μια κανονική χώρα. Αυτή είναι μια παράθεση από μια ανάρτηση στο facebook από ε, μια πηγή παραπληροφόρησης. Βασικός εκδότης πάει συχνά στη Ρωσία, συναντάται με το Ρώσο πρεσβευτή στη Σλοβακία και προσπαθεί να αυξήσει τις δραστηριότητε του φορέα. Ακόμα ε, επεξεργάστηκαν το τιμή της υποψήφια Προέδρου Τζουζάνα Καπούτοβα τότε μέσω Photoshop να φαίνεται πιο ευραία. Το βλέπετε στη φωτογραφία, είναι προφανώς ε, χειραγωγημένη η φωτογραφία. Λοιπόν, Εν ώψη των Ευρωπαϊκών Εκλογών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβαλε διάφορε δράσει, το σχέδιο δράση κατά τη παραπληροφόρηση, ε, το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση ε, και τον κώδικα πρακτική για την αύξηση τη διαφάνεια πολιτικών διαφημίσεων. Πολλοί ανεξάρτητοι ερευνητέ και οργανώσει, παρακολουθώντα την ακαιρεότητα των εκλογών και τα θέματα τη παραπληροφόρηση, βρήκαν ότι υπήρχαν κενά στο σύστημα. Αρκετέ επιχειρήσει ενημέρωση πολύ συχνά ε, τρέχουν παράλληλα από πολιτικούς φορείς της χώρας και από εχθρικές αλλοδαπές ε, δυνάμεις όταν τις παρατηρεί. Είτε αφορά 500 σελίδες του Facebook με ψευδείς πληροφορίες ή διάφορα άλλα αφηγήματα που είναι με αντιευρωπαϊκά ε, μηνύματα της άκρας δεξιάς ε, που απευθύνονται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες ή που προβάλλουν ένα δίκτυο υπέρ του AFD που εντοπίστηκε από δημόσιο κρατικό κανάλι. Και η όλη ιστορία συνεχίζεται. Αυτές οι υποθέσεις είναι η κορυφή του παγόβουνου, διότι βλέποντας περιορισμένους πόρους και τα δεδομένα που έχουμε μπορούμε να εντοπίσουμε μόνο κάποια παραδείγματα, όχι όλα. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς η, αυτός είναι ο σκοπός των επιχειρήσεων, να αλλάξει άποψη του κόσμου, η νοοτροπία του και η πολιτική του προτίμηση. Δυστυχώς, η παραπληροφόρηση και οι σχετικές επιχειρήσεις δεν είναι το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιείται για παρέμβαση στις δημοκρατικέ μας διαδικασίε, Είτε είναι ένα χαλαρό δίκτυο ε, φορέων τη άκρα δεξιά τη Ευρώπη και των ΗΠΑ και διοκτητών προσπαθούν να ανατρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των έσω, δημιουργώντα το κίνημα The Movement υπό την ηγεσία του Steve Bannon, που τον βλέπετε εδώ με τη Μαρίν Λεπέν, ή ρώσικα βρώμικα πετρελοχρήματα που χρηματοδοτούν ιταλικά κόμματα της Ιταλίας όπως το La Liga. Τελικός σκοπός ο ίδιος να ανατρέψουν, να σαμποτάρουν και να επηρεάσουν τις ελεύθερες ε, εκλογές στην Ευρώπη. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ένα κομμάτι άλλο στην εικόνα το παζό. Ε, οι παραστατιωτικές οργανώσεις και διάφορες λέσχες μοτοσυκλέτας. Θα έχετε ακούσει το διαβόητο κλαμπ, τους ε, ε, λύκους της νύχτας, Night Wolves, που παίρνουν εκατομμύρια χρήματα από το πρόεδρο για να κάνουν ε, διαδρομές νίκης ε, από Μόσχα στο Βερολίνο για να τάσουν τη νίκη κατά του φασισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι τιμούμε τις θυσίες που έκανε ο Ερυθρός Στρατός για να μας απο, απελευθερώσει από το φασισμό, αλλά χρησιμοποιεί αυτή την ομάδα την ίδια ευκαιρία, ώστε να διαδώσει φίλο ε, ρωσικά αφηγήματα και εναρμοποίηση τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό ακόμα είναι ότι αυτή η ίδια η ομάδα και τα μέλη αυτής της ομάδας είχαν εμπλακεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, πολεμούσαν στο πλευρό φιλορωσικών αποσυστικών δυνάμεων ε, στο Ντόνετς και, στο, και σε άλλες περιοχές και, εδώ, και στο Ντόμπας. Βλέπετε και στη φωτογραφία. Και μόλις μια χούφτα από εσά ξέρετε ότι αυτή η ομάδα δημιούργησε έδρα ε, στις Ευρώπη στη Σλοβακία, σε ένα μικρό χωριουδάκι, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Πρατισλάβα. Ο ηγέτης του κατάφερε ακόμα να παρουσιαστεί στο Βλαντιμίρ Πούτιν, να συστηθεί στο Βλαντιμίρ Πούτιν και να τον χαιρετήσει διαχειραψίας. Βλέπετε εδώ στη φωτογραφία. Αλλά είμαι σίγουρο ότι αυτό σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τι αστηριότητες στην Ευρώπη. Ναι, δεν θα εκπλήσει κανέναν ότι αυτό εδώ χώρο, αυτή η εγκατάσταση, το Ευρωπαϊκό Αρχηγείο των Night Wolves στη Σλοβακία χρησιμοποιείται σαν τόπο εκπαίδευση και υπάρχει και σκοπευτήριο που χρησιμοποιείται και από άλλε σλοβακικέ παραστατιωτικέ οργανώσει ακόμα και τέτοια οχήματα τάγκ χρησιμοποιούν για να εκπαιδεύονται. Γιατί σα δείχνω αυτά τα, αυτές εικόνες. Ποια είναι η διασύνδεση. Όλες αυτές οι ιδιότητες είναι ένα μικρό κομμάτι μιας ευρύτερης εικόνας του μοσαϊκού, ψηφίδες μοσαϊκού, είτε κυβερνοεπιθέσεις, doxing, ψυχολογικές επιχειρήσεις, ε, πληροφορίες, παραπληροφόρησης, όλα τα άλλα τα στοιχεία, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο στις υβριδικές απειλές όπως αποκαλούνται. Συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία σε μία επιχείρηση μπορείς να πετύχεις στόχους που διαφορετικά δεν ήταν εφικτοί θα ήταν ανέφικτη. Και αυτό αντιμετωπίζουμε. Συντονισμένη, καλοσχεδιασμένη επιχείρηση, καλά χρηματοδοτούμενη από εχθρικέ δυνάμει, κυρίω ρωσικέ δυνάμει, αλλά όλο περισσότερο και από την Κίνα για να ανατρέψουν τι δημοκρατικέ μα κοινωνίε χρησιμοποιώντα βρώμικο χρήμα, παρέμβαση σε εκλογέ, παραπληροφόρηση και κυβέρνοεπιθέσει. Ό,τι θέλετε κάνουν. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ψήφισε ένα ψήφισμα πάνω στο ίδιο θέμα ακριβώς. 4 Οκτωβρίου για την παραπληροφόρηση και παρέμβαση στις εκλογές. Αλλά τα παίρνουμε αυτά όλα αυτά στα σοβαρά. Ένα κοινό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε βρυδικές απειλές και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Στο Ελσίνκι έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για Αριστεία για Ευρυδικές Απειλές στο Ελσίνκι. Αυτό αρκεί, ανταποκρίνεται στην απειλή. Αν κάνουμε μια σύντομη σύγκριση, αν συγκρίνουμε τα ποσά πόρων που διαθέτει η Ρωσική Ομοσπονδία για τα μέσα που είναι κρατικά και τα συγκρίνουμε τα λεφτά αυτά με τους πόρους που διαθέτουν για να εκθέσουμε τα ψευδά, τις ψευδείς ειδήσει, βλέπετε τεράστια διαφορά. 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ επίσημος προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον επόμενο χρόνο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκαλύψουμε τις απάτες και τα ψεύδη. Πώς μπορούμε καν να σκεφτούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες ε, πρακτικές συστάσεις που έχουμε εδώ. Καταρχάς, η προστασία της ακαιρεότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο διαδίκτυο πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα. Να καλύψουμε τα κενά στην νομοθεσία επιχειρηματοδοτήσεως προεκλογική εκστρατεία. Υπάρχουν πολλά κενά. Να εξασφαλίσουμε πλήρη πρόσβαση στι πλατφόρμε κοινωνικών μέσων ε, και για τις διαφημίσεις τι εκλογές για τους ερευνητέ. Να συμπεριλάβουμε τις πολιτικές διαφημίσεις στον έλεγχο που πρέπει να κάνει το Facebook. Να αυξήσουμε σημαντικά τη χρηματοδότηση για δραστηριότητες κατά παραπληροφόρηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρησιμοποιούμε περισσότερα χρήματα. Θα πρέπει να κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αυτό αυτό και να υποστηρίξουμε καινοτόμε λύσει. Και να κλείσω δείχνοντά σα κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν σε μια χώρα με 5 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά μπορεί αυτό να δείξει κάτι και να εμπνευστούν οι άλλες χώρες. Το conspirators.escape για τις διαφημιστικές εταιρείες πώς μπορούν να προστατεύσουν τις πελάτες τους από το να συνδεθούν με ιστοσελίδες κακές και να μειώσουμε τα έσοδα που έχουν αυτές οι κακές ιστοσελίδες. Το Facebook, το Checkbot, ένα ρομπότ επικοινωνιακό, ένα bot που μπορεί να διασταυρώνει τι πληροφορίε, να δει ποιε είναι οι πηγέ, τι γίνεται με τι εικόνε και τι γίνεται με το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Εύληπτο σε τοπική γλώσσα. Εύχριστο. Αν θέλουμε να ενταχθούμε στην πλημμυρίδα, πρέπει να σκεφτούμε καινοτόμα. Θα είχα και ένα βίντεο να παίξω, αλλά μου είπαν ότι θα ήταν βουβό. Οπότε το αφήνω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Thank you. that was good enough, for sure. Φτάνουν αυτά. Πολύ ωραία ήταν. Ε, πάμε τώρα ε, στην τελευταία ομιλήτρια πριν ε, ξεκινήσει η συζήτηση η κυρία Χούγεν Ντούμπελ που εκπροσωπεί την ILGA Europe, ILGA. Έχετε το λόγο για το πολύ 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Κάτρεν Ντούμπελ και είμαι διευθύντρια κοινωνία ΣΥΛΚΑ στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζω ότι έχει περάσει η ώρα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα στην αρχή ότι η ILGA Europe είναι μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης είναι ακρογωνιαίος λήθος κάθε δημοκρατίας. Ε, υπάρχει μεγάλη σύγχυση στη συζήτηση για τη ρητορική μίσους και την ελευθερία του λόγου αυτή τη στιγμή. Και πολύ συχνά η σύγχυση αυτή ε, είναι εσκεμμένη ε, και τη διασπείρουν αυτοί που θέλουν να προβούν σε διακρίσεις και ρητορική μίσους. Σας είπα ότι είναι ακρογωνιαίος λήθος της δημοκρατίας ο ελεύθερος λόγος, αλλά η ρητορική μίσους δεν είναι αυτό. Δεν πρόκειται για ελευθερία της έκφρασης ή διαφορετικές γνώμες. Ε, είναι υποδάβληση ε, μίσους και βίας. Η ρητορική του μίσους, ε, εκούσια ή ακούσια, υποδαβλίζει το μύθος, είναι διακριτικό, είναι κάτι το οποίο δυσφημίζει πρόσωπα ή ομάδες ανάλογα με το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα διάφορα χαρακτηριστικά όταν μιλάμε για τους ΛΟΑΤΚΙ και το μίσος. Ε, η ρητορική μίσους δεν εκφράζει απλώς ιδέες ή διαφορετική άποψη. Προάγει το φόβο, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση προσώπων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ε, παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, ακόμα και απόπειρες αυτοκτονίας. Και μάλιστα όχι μόνο σε πρόσωπα, δεν στοχεύει μόνο άτομα, αλλά και ολόκληρη την κοινότητα. Ε, στον εικονικό κόσμο που, του ίντερνετ το οποίο συζητούμε είναι ακαρία η πληροφορία και όσο ε, προχωρεί αυτό, ανθεί το μίσος. Μίλησαν οι προλαλήσαντες για τον εικονικό κόσμο και τι μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε εκεί το λόγο μίσους. Αυτή τη στιγμή ε, το δίκτυό μας τι βλέπει, ότι αυξάνεται ραγδαία ε, η διχαστική ρητορική, η ρητορική μίσους ε, που οδηγεί πραγματικά σε μίσος και σε βία στην πραγματική ζωή, σε όλη την Ευρώπη, επιτίθεται στον κόσμο και ε, δεν μιλάμε μόνο για δηλώσεις μίσους, ε, αλλά ο κόσμος φοβάται, αισθάνεται ανασφαλής, γιατί αντιμετωπίζει πραγματική βία στην καθημερινή ζωή. Δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο αυτό. Είναι σημαντικό να το θυμίσουμε αυτό. Ε, ε, είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση και πολύ ανησυχητική και πρέπει να το πούμε εδώ. Γιατί ό,τι είναι εικονικό είναι και πραγματικό. Βλέπουμε να αυξάνεται η ρητορική αυτή ε, στις καμπάνιες για δημοψηφίσματα και εκλογές στη δημόσια συζήτηση. Γίνονται από διοπομπέοι ε, τράγοι ε, διάφορες κοινότητες, μειονότητες. Στην Πολωνία πριν από λίγα χρόνια οι πρόσφυγες, φέτος οι ΛΟΑΤΚΙ. Ε, ε, είδαμε την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στην Πολωνία να έρχεται στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με υποδάβληση της βίας. 69 πόλεις και χωριά στην Πολωνία έχουν αυτοανακηρυχθεί ζώνες ελεύθερες από ΛΟΑΤΚΙ αν σκεφτούμε την ιστορία, αυτό είναι μια, ένα καμπανάκι πολύ ανησυχητικό. Ε, βλέπουμε ομοφοβική βία και τρανσφοβική ε, που τεκμηριώνεται από έρευνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι αρχές εβδομάδας του εδώ στη Φιλανδία δημοσιεύτηκε. Τα δικαιώματα των τρανς επίσης ε, ε βάλλονται. Ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει κανονικά την κανονική ζωή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, χρειάζονται ασφάλεια και προστασία από επαγγελματίες. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικό, τους πρώτους έξι μήνες του 2019 αυξήθηκε ο αριθμός των ομοφοβικών ε, εγκλημάτων. Ε, σε σύγκριση με το 2013 μέσα στο πρώτο εξάμεινο είναι περισσότερα εγκλήματα από ό,τι σε όλο το χρόνο. Και αυτό είναι μια τάση που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να υπάρχει διαφορά στο επίπεδο και την κλίμακα της ε, βίας και τον αριθμό των επιθέσεων. Ουσιαστικά, δυστυχώς, είναι μια κοινή απειλή αυτή. αυξάνονται οι πολιτικές δυνάμεις που είναι λαϊκιστικές και εξτρεμιστικές και ε, έχει γίνει πλέον νορμάλ, μπανάλη χρήση αυτών των όρων της βίας λεκτικής που οδηγεί ουσιαστικά και στην πραγματική βία. Επιθέσεις, οι ΛΟΑΤΚΙ δυστυχώς ε, δέχοντο ανέκαθεν. Είναι ε, καθημερινή μας δουλειά αυτή και στις εθνικές οργανώσεις ΛΟΑΤΚΙ αλλά και στην ILGA Europe. Τι έχει αλλάξει όμως και στο προηγούμενο πάνελ ακούσαμε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Για μας τι έχει αλλάξει. Μόνο το 2019 είναι η συχνότητα αυτών των γεγονότων, η σφοδρότητα της βίας. Και τώρα χτυπάνε πάλι σε περιοχές που θεωρούσαμε ότι ήταν ασφαλείς. Δεν υπάρχει μία απάντηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που μας ανησυχεί όλο και περισσότερο. Online ε, είναι διεθνής η δράση με δράστες και θύματα παντού και οι πλατφόρμες έχουν ε, έδρα αλλού και ο σερβερ αλλού πάλι. Ε, υπάρχει ένα νομικό, πρακτικό και πολιτικό πλαίσιο πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχει σαφήνεια για το ποια χώρα ε, ε, θα πρέπει να διώξει, ποια είναι η δικαιοδοσία και πώς θα υποστηριχθούν τα θύματα. Πολύ συχνά ακούμε στη συζήτηση ότι ό,τι ότι είναι παράνομο στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική ζωή, θα πρέπει να είναι παράνομο και ηλεκτρονικά. Αν δούμε όμως ε, τη φοβία και το μίσος των ΛΟΑΤ από εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Σήμερα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που να επιβάλλει σε όλα τα κράτη-μέλη να ποινικοποιούν τα εγκλήματα μίσους ή τη ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Η βασική νομοθεσία στην Ευρώπη είναι ε, μια απόφαση πλαίσιο του 2008 του Συμβουλίου που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να ε, τιμωρούν τα κίνητρα όταν είναι ξενοφοβικά, ρατσιστικά κτλ και ε, όταν υπάρχει άρνηση ή ε, υποτίμηση του ολοκαυτώματος. Ε, ωστόσο για τους ΛΟΑΤΚΙ κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Σε εθνικό επίπεδο, επίπεδο, κράτη-μέλη της Ένωσης δεν έχουν βάλει στην νομοθεσία ρητορική μίσους το θέμα αυτό του γενετήσου προσανατολισμού, ούτε της Ταυτότητα του φύλου. 15 κράτη-μέλη και κανένα κράτος δεν ε, ασχολείται με τους μεσοφιλικούς. Η νομική προστασία των δικαιωμάτων, ΛΟΑΤΚΙ, είναι κάτι που μετράμε και τσεκάρουμε. Ε, εσείς μπορείτε να το βρείτε για ποιες χώρες πρόκειται. Η νομοθεσία παράγει κουλτούρα, πολιτισμό και δείχνει τι κοινωνία θέλουμε. Και αν συζητούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τη ρητορική μίσου online και offline, πρέπει να βλέπουμε πάντα και το νομοθετικό πλαίσιο. Αν μια κυβέρνηση ε, συμπεριλαμβάνει αυτά στη νομοθεσία ε, για τη ρητορική μίσου ε, λαμβάνει θέση απέναντι σε αυτό το μίσος. Και επίσης επιτρέπει αυτό συνέχεια παρακολούθηση και σωστή δίωξη. Θα ήθελα μόνο να σας αφέρω ακόμα ένα παράδειγμα. Ακούσαμε για την πολωνική τηλεόραση προηγουμένως. Άλλο παράδειγμα, ε, το 2018 πριν το δημοψήφισμα για τον ορισμό της οικογένειας στη Ρουμανία, μια διαφήμιση ε, ε, του PSD που μιλούσε για την ισότητα ε, και έλεγε ότι όταν παντρεύεσαι άτομο του ιδίου φίλου είναι σαν να παντρεύεσαι ένα φυτό, είναι ένα αντικείμενο και χάνεις τη λογική σου δηλαδή και την ηθική σου. Ε, αυτό σημαίνει υποσυνείδητα ή ε, εννοεί ότι οι ΛΟΑΤΚΙ είναι κατώτερα άτομα και είναι μια απειλή ε, που προάγει την ρητορική μίσους και το κλίμα η ρουμανική μας οργάνωση έκανε καταγγελία στη ρουμανική κυβέρνηση στις αρμόδιες αρχές που δεν έδωσαν συνέχεια. Ε, ε, όλοι λοιπόν οι, άνθρωποι αυτοί οι ΛΟΑΤ όσοι έχουν διαφορά για λόγους φίλου και, και για διάφορους άλλους λόγους το έχουν ζήσει στο πετσί τους. Τι ε, μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Νομική προστασία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. E Υπάρχει μια σύσταση για το παράνομο περιεχόμενο. Υπάρχουν διάφορες μορφές παράνομου περιεχομένου και διάφοροι τρόποι ε, να αντιμετωπιστεί αυτό. Μπορεί να υπάρξουν και στοχευμένα νομοθετικά μέτρα. Αλλά δεν, δεν αναφέρονται τα κίνητρα πάντα ρητά. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πολιτική ηγεσία αντιμετώπιση του ίσους και να προσέξουμε να μην πούμε σε μια ψευδή συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία της έκφρασης και να διαφυλάσσεται. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι ε, υπάρχει κατάχρηση από διάφορες ε, οργανώσεις που θέλουν να κάνουν διακρίσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο το ΛΟΑΤΚΙ, αλλά κατά των γυναικών, των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων μειονοτήτων. Σε ό,τι αφορά το μίσος online βλέπουμε ε, ένα ψηφιδωτό λύσεων γίνονται συζητήσεις με εσά, τους εκλεγμένους εκπροσώπους, ε, με άλλους εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές και ε, οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων για να εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ε, εκπαίδευση για το διαδίκτυο είναι πραγματικά κλειδί σε αυτές τις συζητήσεις. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολικά δραματικά αυτά που λέω, ακούγοντας και τους άλλους ε, ε, ομιλητές, να πούμε ότι πραγματικά η κατάσταση είναι ανησυχητική, αυξάνεται το μίσος. Είμαστε τώρα σε ένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να υπάρξει πολιτική ηγεσία και από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμο για να ε, σταματήσει αυτό το μίσος και να ε, εκπέμψουμε και πολιτικά αλλά και νομοθετικά μηνύματα για να καταπολεμήσουμε το μίσος εντός και εκτός του διαδικτύου. Σας ε, ευχαριστούμε. Θα κάνουν οι βουλευτές ερωτήσεις στους ομιλητές. Όσοι θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Μένατε χειρός και εμείς θα σημειώσουμε. Okay, you take note. Pelletier and Tang. Yeah, but I understand that the, uh, you also too. You want to? I understand that the Commission would also. Από ό,τι καταλαβαίνω και η Κομισιόν θα ήθελε να σχολιάσει στη συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μια σύντομη δήλωση, σας ευχαριστούμε έτσι ώστε να γλιτώσουμε χρόνο για τους βουλευτές. Γιατί βλέπω ότι είναι και περισσότεροι ζητούν το λόγο. Μπορείτε να είστε σύντομος, παρακαλώ, ή σύντομοι. Ευχαριστώ για το θέμα της ρητορικής μίσους και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για την παραπληροφόρηση. Ακούσαμε από τους ομιλητές ότι η ρητορική μίσους είναι αυξανόμενο πρόβλημα και γίνεται κάτι που κανονικοποιείται. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε την ιστορία μας και να είμαστε Προσεκτική να επαγρυπνούμε γιατί στην πυραμίδα του μίσους όταν έχουμε ρητορική μίσου στην κοινωνία ήδη αυτό είναι ένα ε, σημάδι προειδοποίησης που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη ρητορική μίσους. Έχουμε την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία υποχρεώνει τα να ποινικοποιήσουν ε, πράξεις ε, δημόσιας παρακίνησης ε, σε βία και μίσος βάσει συγκεκριμένων προστατευόμενων χαρακτηριστικών. Φυσικά, αυτό το είδος του λόγου θα πρέπει να διαχωριστεί από το λόγο που ε, όσο ε, και αν προσβάλλει, προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα, όχι με το ποινικό δίκαιο ή με την ε, αφαίρεση των λόγων αυτών από τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνική δικτύωσης ή νόμοι είναι καλοί μόνο αν εφαρμόζονται αποτελεσματικά επί τόπου. Έτσι λοιπόν Οι Κομισιόν έχει ιδιαίτερα ενεργά συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αποτελεσματικές έρευνες και επιβολής της νομοθεσίας τόπου. Και αυτό το κάνουμε στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επίπεδου για το ρατσισμό και την ξενοφοβία και άλλες μορφές μεσαλλοδοξίας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο συνεκτικοί στο έργο μας. Ωστόσο, δεδομένου ότι το περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει τόσο σημαντικό φόρουμ για παράνομη ρητορική μίσους. Αυτές οι προσπάθειες να βεβαιώσουμε ότι η ρητορική μίσους ε, ε, ερευνάται και διώκεται αποτελεσματικά πρέπει να συμπληρωθεί με δράσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ε, κάνουν και αυτές αυτό που τους αναλογεί για να διασφαλίσουν ότι ε, η ρητορική μίσος που το κοινοποιείται ε, αφαιρείται για τον κώδικα δοντολογίας του 2016 που υιοθετήθηκε από το Facebook, το Twitter, το YouTube και τη Microsoft οι εταιρείε δεσμεύτηκαν ε, να δρουν εγκαίρους εντός 24 ώρου κατόπιν κοινοποίηση παράνομης ρητορική μίσους και να αξιολογούν αυτές τις κοινοποίησει και να αφαιρούν το περιεχόμενο αν θεωρείται παράνομο. Εμείς ε, συνεργαστήκαμε με την κοινωνία των πολιτών για να δοκιμάσουμε πώς λειτουργεί ο κώδικας δεντολογίας στην πράξη. Η παρακολούθηση που κάναμε μας δείχνει συνεχή πρόοδο. Έχουμε συνεχή αύξηση στα ποσοστά αφαίρεση. Η τελευταία αξιολόγηση που δημιουργήθηκε το 2019 μας έδειξε ότι οι εταιρείε αφαιρούν τώρα το 70% των κοινοποιήσεων, του λόγου που κοινοποιείται σε αυτούς σε σύγκριση με το 28% το 2016. Αλλά νομίζω τώρα ότι το πιο πολύτιμο αποτέλεσμα του κώδικα είναι ότι έχει οδήγησε σε μια συνεργατική προσέγγιση μεταξύ κοινωνίας των πολιτών, των πλατφορμών και των κρατών μελών. Και θέλουμε να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οπότε κατάλαβα ότι υπήρχε και δεύτερος εκπρόσωπος Κομισιόν που θέλει το λόγο κάποιε παρατηρήσει για τη ρητορική μίσου, αλλά μην με κρηγορείτε, παρακαλώ. Γιατί έχουμε ένα κατάλογο από 15 βουλευτέ. Και σήμερα το πρωί μείναμε στην αίθουσα αυτή για πάνω από, μία, από μισή ώρα. Και μα περίμεναν συντονιστέ. Και μείναμε και χωρί διερμηνία για πάνω από μισή ώρα. Δεν θα πρέπει να συμβεί και απόψε. Μην με παρακαλώ. Απλώ θα κάνω μια επικαιροποίηση για τον κώδικα πρακτικής και τη σχετική πρόοδο για την παραπληροφόρηση. Ο κώδικα. Ε, τώρα είναι ενό έτου, ε, και έχουμε μία προσπάθεια κανονιστική που έχει υπογραφεί από τις κύριες πλατφόρμες online και από τους εκπροσώπους της ε, διαφημιστικής βιομηχανίας. Η Κομισιόν τώρα είναι στη διαδικασία του να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει λάβει χώρα. Η αυτοξιολόγηση που έγινε από τα υπογράφοντα μέρη έδειξε ότι ο κώδικας ε, ε, οδήγησε σε μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις ε, πολιτικές των πλατφορμών για το κατεβέσμα της πληροφόρησης μας ενημέρωσαν για τις δράσεις που έχουν λάβει για να περιορίσουν τη δυνατότητα παρέμβασης από κακόβουλους δράστες όμως παραμένει αναγκαιότητα να συμμετέχει όλη η κοινότητα η για κυριότητα των υπηρεσιών και ε, κάποιες λόγω δοσίας αλλά και διαφανείς διαφημίσεις χρειάζονται. Αυτό οφείλεται και στην παρακολούθηση των διαμέσων που γίνεται κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών. Η ενδυνάμωση των χρηστών ε, είναι το μέσο όπου ε, υπολείπεται ε, ο κώδικας, η εφαρμογή του κώδικα. Ε, δεν ε, έχουν εφαρμοστεί παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολιτικές. Ένα ε, παράδειγμα αυτής της είναι το fact-checking, ένα από τα κύρια εκκρεμή θέματα παραμένει η πρόσβαση στα online δεδομένα για δημόσιο έλεγχο. Βασιζόμαστε μόνο στις εκθέσεις της αυτοξιολόγηση αυτή τη στιγμή και για ερευνητικού σκοπούς, γιατί οι πλατφόρμες θα πρέπει να αυξήσουν την προσπαθία του στο θέμα αυτό. Αναμένουμε πρόοδο μέσω του ε, επόμενου παρατηρητηρίου για τα ψηφιακά μίντια που υλοποιεί η Ευρώπη μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility. Δεν ε, θα δώσει το παρατηρητήριο μέσα μόνο για μια πολυτεμιακή κοινότητα να αυξήσει την ανάλυση της ε, εκστρατείας παραπληροφόρησης, αλλά δημιουργούμε και τις συνθήκες για να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα βάσει των κανόνων της προστασίας των δεδομένων. Ένας τρόπος που θα έχει σχεδιαστεί σωστά για την πρόσβαση στα δεδομένα θα βοηθήσει την την ε, ε, πολιτική των ε, πλατφόρμων και θα απαντήσει στη συγκεκριμένη ανάγκη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η αξιολόγηση της Κομισιόν θα συνεχιστεί του επόμενου μήνε, Αυτή η αξιολόγηση θα αποτιμήσει τη δουλειά που έχει γίνει από ένα εξάρτητο τρίτο μέρος που θα έχει διοριστεί από τους υπογράφοντες του κώδικα, από μια μόνιμη επιτροπή ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια έκθεση που από τις αρχές έργα και την έκθεση της ε, Κομισιόν για τις ευρωεκλογέ του 19. Μια πλήρης αξιολόγηση θα είναι έτοιμη αρχές του 2020 και αν δεν είναι αποτελεσ... ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, η Κομισιόν μπορεί να προτείνει νέα μέτρα και κανονιστικής ε, φύσεως. Βέβαια, έχουμε πάντοτε κατά νου την προστασία της ελευθερίας τη έκφρασης. Σας λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα έχουμε 15 ε, μέλη, 4 ε, μέλη του πάνελ και πρέπει να απαντήσουν. Παρακαλώ κάντε τις ερωτήσεις σας έτσι ώστε να μπορούν να απαντηθούν. Ένα λεπτό για να μιλήσετε όλοι. Okay, we get started. The first Πάμε. Ο, ο κύριος Ρουίθ Ντεβέσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας. Εγώ δεν έχω τόσο πολλή ερώτηση. Μάλλον ε, μια σκέψη θέλω να μοιραστώ μαζί σας μετά από αυτά που ακούσαμε. Όλες οι παρουσιάσεις τονίζουν ε, ε, και φωτίζουν τις διάφορες διαστάσεις του φαινομένου που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Παραπληροφόρηση, ξένες επεμβάσεις σε διαβουλεύσεις σε διαδικασίες λήψης απόφασης, σε εκλογές και ρητορική μίσους. Όλα αυτά είναι θέματα και δυναμικές που συνδέονται. με την αρνητική ε, χρειά. Αυτοί που χρησιμοποιούν καμπάνιες παραπληροφόρησης, καμιά φορά ε, προάγουν και τη ρητορική μίσου στην απόρριψη του διαφορετικού. Πού βρισκόμαστε, έχουμε μια πρόκληση απέναντί μας ως θεσμικό όργανο και ως βουλευτές να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να στρώσουμε μια πολυδιάστατη ολιστική στρατηγική από την προστασία της ε, διερευνητικής δημοσιογραφίας, ερευνητικής μάλλον, ε, ε, καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και ελευθεροτυπία. Έλεγε προηγουμένως η κυρία Φόξ ότι είναι κατά της επίσημης αλήθειας. Καλά, μπορεί κάποιος να έχει ελεύθερη γνώμη και άποψη στα πλαίσια του νόμου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό που δεν μπορεί να έχει είναι να επιτρέπει να εφευρίσκουμε ειδήσει ε, γεγονότα που δεν συνέβησαν. Ευχαριστώ, η κυρία Ρίβα. Ε, καλησπέρα σας. Θα μιλήσω για ένα θέμα που ακούσαμε από τον κύριο Μήλο προηγουμένως πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτό το αυταρχικό καθεστώς. Στις 18 Οκτωβρίου η χωροφυλακή μετά από ε, εντολή δικαστική ε, ε, ζήτησε από την Microsoft να κλείσει μια ιστοσελίδα του Tsunami Democratic στην ε, Καταλωνία. Ε, μα δεν μπορείς να κατηγορείς για τρομοκρατία ανθρώπους που διαμαρτύρονται θεμητά η ελευθερία της έκφρασης και ε, του διαδηλώνει. Η Διεθνής Αμνηστία λέει ότι η Ισπανία χρησιμοποιεί με κακό τρόπο τον ποινικό κώδικα και ε, κυνηγάει αντιφρονούντες ε, και ε, τους επιβάλλει λογοκρισία χαρακτηρίζοντάς τους τρομοκράτες. Και όχι μόνο διαδηλωτές αλλά και καλλιτέχνες, ε, τραγουδιστές και τα μόλις η κυβέρνηση, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ ενέκρινε διάταγμα νόμο που θα επιτρέπει χωρίς δικαστική εντολή για λόγους δημόσιας τάξης η εκτελεστική εξουσία να κλείνει στο σελίδες. Αυτό ε, ανοίγει ένα προηγούμενο πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι πιστεύετε ε, για αυτά τα πράγματα. Ε, κυβερνήσεις χωρί εντολή δικαστική να κλείνουν ε, ε, στο σελίδες. Και τι θα συστήνατε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύουν με τρόπο αποτελεσματικό τους πολίτες από αυτές τις επιθέσεις στην ελευθερία της έκφρασης. Ευχαριστώ. Κυρία Αδαμόβιτ, ευχαριστώ πολύ τα μέλη του πάνελ για τις παρουσιάσεις και τα παραδείγματα που παρέθεσαν. Έχω μια ερώτηση για την κυρία Μαζούρκεβιτ. Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν οι ΜΚΟ στην πάλη κατά της παραπληροφόρησης και των λόγων μίσους, τι μπορεί να γίνει για να ενισχυθεί η λειτουργία των λόγω φορέων, τι μπορεί να βοηθήσει τις ΜΚΟ για να πετύχουν κάποιες συνεργασίες με πρωτο... μαζί με τις πρωτοβουλίες των πολιτών. ΜΚΟ με, με πρωτοβουλίες πολιτών και πώς μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού της παραπληροφόρησης. Κύριε Κέλλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τους υπευθύνους των ΜΚΟ που μας παρουσίασαν τις θέσεις τους. Σας χαιρετίζω και αναγνωρίζω την προσπάθεια που κάνετε, τις δράσεις που καταβάλλετε κατά των λόγων μίσους. Πρέπει να πω ότι αυτή η ελευθερία του λόγου έχει άρει φράγματα, επιτρέπει ε, τελικά όμως ομιλίες απαράδεκτες και ταχεία διάδοση κατά τον ΛΟΑΤΚΙ, κατά κάποιων των άλλων και υπενθυμίζει τις πιο μαύρες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας αυτό το φαινόμενο. Από την πλευρά μου είμαι πολύ θετική για μεγαλύτερη ευθύνη των πλατφορμών να αφαιρούν αυτά τα περιεχόμενα τάχιστα. Ποια είναι η άποψή σα μεταξύ ελευθερία έκφραση και ταχεία απόσυσης των αναρτήσεων. Ποια είναι η ισορροπία. Στην Ισπανία έχετε κάποιε αναξαρτησίε σχετικά με το ποιο έχει την ευθύνη, ποιο κατευθύνει αυτή την απόσυση. Μπορεί να γίνει κάτι υποχρεωτικό, αλλά χρειάζεται και κάποιο αντιστάθμισμα, κάποιο έλεγχο, κάποια υποπτία. στι ευρωπαϊκέ εκλογέ, άκουσα πολλού πολίτε, οι οποίοι είχαν επίγνωση της χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης και έδειχναν ότι δεν πιστεύουν πλέον στην εκλογική διαδικασία και αμφισβητούν και τα αποτελέσματα των εκλογών μου λέγανε είναι προδιαγεγραμμένα, χειραγώγηση έχει γίνει κλπ. Έχετε κάποια σχετικά μηνύματα. Ποια είναι η απόψή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόξ. Κυρία Φόξ, έχετε το λόγο. Μισώ τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και την αλαζονία κατά των εργαζομένων, αυθαίρε τους πολιτικούς. Έχω πολύ μίσος μέσα μου. Πρέπει να με φημώσουν. Λυπάμαι, φοβάμαι ότι οι μεγαλύτερε απειλέ για την ελευθερία του λόγου είναι η νομοθεσία κατά των λόγων μίσους. Φημώνει την νόμιμη έκφραση του λόγου, κανονικά η νομιμή, νόμιμη έκφραση των αντιπάλων σου. Ποιο αποφασίζει τι είναι μίσος, ένας από τους ομιλητές της πλατφόρμας το είπε και είχε δίκιο κυρία ότι η το κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ ε, αντιμετωπίζει με τοξική ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει ότι οι νόμιες ανησυχίες που εκφράζουν οι λεσβίες και οι φεμινίστριες που ανησυχούν για κάποιες θεότητες άλλων των φιλομεταβατικών απαγορεύεται να συμμετέχουν στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Τους κυνηγάει αστυνομία και κατηγορούνται και αυτό οδηγεί τελικά σε επιθέσεις σε κάθε είδους ανθρώπους όπω τα μέσα ενημέρωση και του δημοσιογράφου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθεροτυπία και ελευθερία λόγου και μετά να επιχειρηματολογούμε οι υπέρ μέτρων που φημώνουν το λόγο. Αυτό είναι κατά τι προσπάθειε για πιο μεγαλύτερη ελευθερία λόγου και ανταλλαγή επιχειρηματών. Και η παρακίνηση δεν είναι ε, κάτι αυτόματο. Εγώ, μα ακούτε να μιλάω, δεν συμφωνείτε αυτομάτω με μένα. Δεν του λένε το άλλο να πηδήξει από τον κρεμό και πηδάει απαραίτητα. Δεν θα πρέπει η παρακίνηση να θεωρείται ότι είναι ένα αίτιο μέσω του οποίου μπορούμε από την πίσω πόρτα να επιφέρουμε φήμωση στην ελευθερία της έκφρασης. Ευχαριστώ κύριο Μπίσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίλτσικ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Έκαναν έξοχες παρουσιάσεις. Σαφέστατα τις παρουσιάσεις ήταν ότι η διάδοση της παραπληροφόρησης δεν είναι κάτι που θα εξαφανιστεί εφάπαξ φαινόμενο, αλλά είναι συστηματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστηματικό τρόπο. Εξού και η ερώτησή μου. Προσεκτικά υποβάλλετε συστάσεις. Μπορείτε να είστε πιο τολμηροί. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς που θεσπίζουμε νομοθεσία, κατά την άποψή σας διδατορικοί κώδικες και πρακτικές είναι χρήσιμα στοιχεία, αλλά έχουν και περιορισμούς. Ερώτηση προς όλους. Πώς βλέπετε την καλύτερη δυνατή λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ιδανικά. Δεν είναι ένα αυθαίρετο πρόβλημα, αλλά είναι ένα θέμα συστημικό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε μέσω πολιτικής αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Τα παραδείγματα που ακούσαμε πραγματικά είναι τρομακτικά. Όμως, εδώ μπορεί να βρισκόμαστε ενίοτε μεταξύ ελεύθερου λόγου και ρητορικής μίσου. Και ακούσαμε το θέμα της αυτοξιολόγησης από τις πλατφόρμες, ε, δεδομένα που δεν ε, ε, τα μοιράζονται και που πρέπει και ξέρουμε ότι οι αλγόριθμοι επίσης λειτουργούν προς το να τραβούν την προσοχή, δηλαδή ε, τελικά διαδίδεται η ρητορική μίσους και αυτό είναι μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου των πλατφορμών δεν θα ήθελα να σιωπάτε γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι η διάχυση της ιστορικής μίσους online είναι πολύ σημαντικό, καθώς αυτό μεγενθύνεται και επιροδοτεί ε, και ε, offline, εκτός του διαδικτύου, τη ρητορική μίσους. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να περιορίσουμε τις πλατφόρμες και να δώσουμε νέες κατευθύνσεις στον τρόπο εργασίας τους. Θέλουμε να ακούσουμε τα σχολιά σας γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σπράιερ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές ε, για την ομιλία τους ε, και είναι σαφές ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και της ανοιχτής κοινωνίας βρίσκονται υπό πίεση και επίθεση. Ακόμη και ε, η εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς απειλείται. Ακούσαμε τον κύριο Μίλο και τον κύριο Ναράχο και μου άρεσαν αυτά που πρότειναν, αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις αξίες μας. Κάποιες λύσεις που προτάθηκαν από άλλους φορείς είναι προβληματικές νομίζω. Δεν θα πρέπει η βιομηχανία, ο κλάδος να αποφασίσει για το βαθμό της ελευθερίας έκφρασης ε, online. Αυτό είναι ένα δημόσιο θέμα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με ένα άλλο επίμαχο θέμα, το είναι ανώνυμη ρητορική είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τις μειονότητες και τις μειονοτικές απόψεις και τα θύματα της παρενόχλησης να μπορούν να συζητούν ανώνυμα χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Όμως κάποιοι άλλοι λένε ότι κάθε ε, ρητορική, κάθε λόγος ε, θα πρέπει να μπορεί να ταυτοποιηθεί. Και ξέρετε ότι υπάρχει στην Αυστρία κάποια σχετική νομοθεσία ε, τώρα, ε, έχουμε δει ότι οι λογαριασμοί πραγματικά ονόματα χρησιμοποιούνται για να διαδίδουν ακόμα και περισσότερο μίσος ε, online από τους ανώνυμους λογαριασμούς. Ποιε είναι οι απόψεις σας για το θέμα αυτό? Θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα σε ανώνυμο λόγο? Ή πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει? Να ευχαριστώ κύριο Βάιμερς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ θέλουμε να συζητήσουμε τις ψευδείς ειδήσει. Θα θυμόσαστε όταν η δική μου χώρα είχε περιγράψει κάποιες γειτονιές σαν περιοχές όπου δεν μπορεί να πάει κανείς. Τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες ότι έπρεπε να φοράνε λεξίσφαιρα γυλαίκα οι οδηγοί νοσοκομιακών ασθενοφόρων. Υπάρχουν επικίνδυνες περιοχές στην Σουηδία που αποκαλούνται απαγορευμένες ζώνες, no-go zones. Και το Συνδικάτο των Ασθενοφόρων λέει ότι υπάρχουν τέτοιες περιοχές, ότι για μας ισχύει. Είναι απαγορευμένη περιοχή, η τάδε η περιοχή. Και οδηγίε είναι να μην πηγαίνουμε σε αυτέ τι επικίνδυνε περιοχέ και να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνε καταστάσει. Έχουμε λοιπόν μία δήλωση του Συνδικάτου των ε, Οδηγών Ασθενοφόρων. Αυτό τι είναι, ψευδή είδηση. Δεν είναι μεγάλη ευθύνη εμείς εδώ να καθόμαστε, εδώ στο Κοινοβούλιο, μακριά και κάποιες δηλώσεις να τις αποκαλούμε ψευδείς ειδήσει. Υπάρχουν τέτοιες περιοχές απαγορευμένες επικίνδυνες πολύ στη Σουηδία, όπου εκρήγνονται, και διάφορες βόμβες. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριο Σούρχρικ. Ε, θα ήθελα να ε, σας μιλήσω για τον Ντάνιελ ε, Μούλερ, που δεν έχει γεννηθεί στη Σλοβακία, δουλεύει για την Globsec, που χρηματοδοτείται από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών απευθείας. Και λίγο περίεργο μου φαίνεται που μιλάει για τις ξένες επεμβάσεις σε εκλογές ή σε κράτη. Ε, πρέπει εγώ να ε, υπερασπιστώ τη Σλοβακία και του Σλοβάκους. Είναι ψεύδι αυτά που λέει. Ούτε αντισημίτες είναι οι Σλοβάκοι, ούτε εξτρεμιστές. Ε, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άνθρωποι καλοί, αξιοπρεπείς, ε, εργαζόμενοι σκληρά. Μα πώς είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος εδώ στο κοινοβούλιο να λέει τέτοια πράγματα. Το πρόβλημα που έχουμε στη Σλοβακία είναι με κάτι εξτρεμιστές πολιτικούς, φιλελεύθερους υποτίθεται, που θέλουν να φημώσουν κάποιους άλλους με πρόφαση ε, τον αγώνα κατά των εξτρεμιστών. Κυρία Τούν, ευχαριστώ. Εγώ χάρηκα που γνώρισα τον κύριο Μήλο, που είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής και εργαζόμενος ε, σκληρά και μας έκανε μια φανταστική παρουσίαση. Ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά ακούγονται ωραία και καλά, συνεχιζόμενη πρόοδος, ε, όλο και περισσότερο συμβαλώμενα μέρη υπογράφονται, ξέρω εγώ, αλλά όλο και περισσότερα fake news βλέπουμε, ε, απειλές, ψευδείς ειδήσει και μίσος στις πλατφόρμες. Ποιος φέρει την ευθύνη, οι πλατφόρμες, αυτό είναι το θέμα. Ε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το Facebook, για παράδειγμα, δεν δίνει τις πληροφορίες σε σχέση με τους ανώνυμους λογαριασμούς που ρωτήσατε. Αρνείται να δίνει πληροφορίες στο Facebook και δεδομένα και στοιχεία για τους συντάκτες αυτών των απειλών ακόμα ε, ε, και αν το ζητάει η εισαγγελία. Δηλαδή, ε, πραγματικά υπάρχει κάποιο όριο. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν μπορούμε να φτιάχνουμε ασπίδες αντιπυραυλικές για πυράβλους που μας απειλούν. Γιατί δεν μπορούμε να εργαστούμε όλοι για να φτιάξουμε μια αντιπυραυλική ασπίδα ε, του πυράβλου των fake news και του μίσους που σιγά σιγά απειλεί και τη ζωή την ίδια κάποιων ανθρώπων και σίγουρα τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο πρέπει να φτιάξουμε αυτό το checkpoint που ανέφερε ο κύριος Μήλο, που δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί αυτό το φυλάκι, ας πούμε, θα ήταν μια καλή αρχή. Ο πρόεδρος, δεν νομίζω να ξέχασα κανέναν. Α, η κυρία Ίνσε, ε, ένα λεπτό. Και μετά να δώσουμε λίγο και το λόγο για τις απαντήσεις. Θα πάω απευθείας στην ερώτησή μου. Χρειάζεται αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο ε, για να βελτιωθεί η νομοθεσία και να μην έχουμε ε, ρητορική μίσους για να διώκονται τα ρατσιστικά εγκλήματα. Μιλώ για το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπατε ότι είναι μόνο ε, μία απόφαση πλαίσιο ε, για το πώς θα διωχθούν ποινικά τέτοια φαινόμενα. Επανέρχομαι στο πάνελ και παρακαλώ. ότι έχετε υπόψη σας ότι η συζήτηση δεν τελειώνει εδώ. Απλώς απαντήστε στις ερωτήσεις. Δεν είναι τα καταληκτικά σχόλια αυτά όλων των εποχών. Το συντομότερο δυνατό, παρακαλώ. Η ε, κυρία Μαρκουσέβιτς. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, να απαντήσω στο τι πρέπει να κάνει η κοινωνία των πολιτών. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Μίλο εδώ, γιατί πιστεύω ότι αφενός ε, βλέπουμε ότι υπάρχει όλος ο λαϊκισμός, όλοι οι λαϊκιστές που εργάζονται μαζί και θα πρέπει και εμείς να συγκεντρωθούμε στην πλευρά μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και να ελέγξουμε τι συμβαίνει με την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την κοινωνία των πολιτών, αλλά και για τους πολίτες, αλλά και τους πολιτικούς. Πιστεύω ότι είμαστε πιο ισχυροί, ενωμένοι και αν μπορέσουμε να εργαστούμε χρησιμοποιώντα τι ικανότητέ μας ε, και χρησιμοποιήσουμε όσα έχουν ήδη παραχθεί, τότε μπορούμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Πιστεύω κάθετα ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς ε, ως νομοθέτες είναι να φέρετε περισσότερη χρηματοδότηση στον τομέα αυτό. Υπόθηκε, αλλά είναι ζωτικό όχι μόνο η Ρωσία αλλά και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται στο θέμα της παραπληροφόρησης ρίχνουν πάρα πολλά χρήματα. Το βλέπουμε αυτό στο διαδίκτυο και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Τώρα, η απάντησή μου για το τι μπορούμε να κάνουμε είναι συνεργασία, ενδυνάμωση της συνεργασίας, επικοινωνία, γιατί ξεχνάμε το θέμα της επικοινωνίας Συχνά γράφουμε πολλές μεγάλες εκθέσεις και λέμε στους ανθρώπους ότι θα πρέπει να διαβάζουν άρθρα ή βιβλία αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να κοινοποιούμε τα μηνύματα με απλό τρόπο και να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, να έχουμε μια απλή επικοινωνία που να έχει απεύθυνση στους πολίτες. Χρειαζόμαστε εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Πρέπει να δούμε ευρύτερα την όλη εικόνα και να απευθυνόμαστε σε διάφορες ομάδες ε, και να δούμε τι δουλειά δίνεται για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Και φυσικά εκπαίδευση είναι ζωτική, είναι βασική, γιατί οι άνθρωποι τείνουν περισσότερο στην περιπληροφόρηση όταν ε, δεν έχουν συνέστηση. Και επίσης, δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις πληροφορίες εκεί, αλλά οι εξτρατείες της πληροφόρησης για την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους είναι ζωτική σημασία. Δεν νομίζω ότι ε, η ρητορική μίσους είναι το ίδιο σαν να μιλάμε για την ελευθερία τύπου. Ήδη έχουμε ποινικοποιήσει τη ρητορική μίσους offline, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και online. Παραδείγματο χάρη, δεν ποινικοποιείται η ρητορική μίσου στην Πολωνία κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Ε, έτσι λοιπόν, άνθρωποι που προσβάλλονται από τη ρητορική μίσου ε, δεν ποινικοποιούνται. Και αυτή η νομοθεσία είναι πολύ σημαντική εδώ. Επίσης μιλήσαμε πολύ για μίσος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλώνει την κοινωνία των μίσος. Δεν ξέρουμε πού θα πάει και πού θα καταλήξει. Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε. Και αν δεν δώσουμε προσοχή και δράσουμε τώρα, δεν ξέρουμε που θα βρισκόμαστε σε ένα-δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ναράγχο. Ναι, σε σχέση με την κατάσταση στην ε, Καταλωνία, ήδη μιλήσαμε για το τσουνάμι δημοκράτικο. Ε, υπήρξαν κάποιες αποδείξεις ε, και γι' αυτό έγινε η σχετική έρευνα και θα ήθελα να δω αυτή την έρευνα γιατί αυτό που είδα είναι ειρηνικά κινήματα υπήρξαν ε, κάποια φαινόμενα όπως και σε άλλες διαμαρτυρίες κάποιες βίες πράξεις όμως δεν, αν δεν είναι τρομοκρατία τότε τι ερευνά που πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα Επίσης, ε, δεν ε, έχω εξετάσει ε, το θέμα εγώ ίδιος, αλλά έχουμε έμπιστες πηγές στην Ισπανία για το ότι αποτελεί δικαστής αυτός άλλη απειλή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα για το πώς θα εξελίξουμε τις ΜΚΟ, καλωσορίζουμε, να τις καλωσορίζουμε στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε την ικανότητα να δράσουμε. Εγώ έχω τον πάτσι μου και έρχομαι εδώ συχνά, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, δεν ισχύει αυτό για πολλούς άλλους. Φέτος ε, φέραμε 17 ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη για να δράσουν κατά τις οδηγίες για το copyright και στη συνέχεια μας κατηγόρησε ότι παραπληροφορούμε τους ευρωβουλευτές. Ε, νομίζω ότι είναι κακή ιδέα να μην συμμετέχουν οι άνθρωποι στις πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ερώτηση, κυρία Σκέλερ, τι να κάνουμε. Δεν λειτουργούν τα φίλτρα. Έτσι λοιπόν, το να ανεβάζουμε φίλτρα δεν δουλεύει ε, ίσως ε, θα χρειαζόταν ένας ε, μηχανισμός ε, που να προκρίνει σε διάφορες δράσεις ανάλογα με τα διάφορα είδη περιεχομένου. Ίσως αυτό να ήταν μια καλή ιδέα στην μελλοντική νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Επίσης πρέπει να επιτεθούμε στο επιχειρηματικό μοντέλο. Νομίζω είστε σε θέση τώρα για να υιοθετηθεί ο κανονισμός από την γαλλική κυβέρνηση για το e-privacy, γιατί μπλοκάρεται εδώ και δύο χρόνια και κατόπιν να εφαρμοστεί ο, κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των δεδομένων ε, και θα πρέπει να παρακολουθεί και το τι συμβαίνει ε, ο EDPS. Τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η απειλή ε, το να απειλούνται online διάφορα άτομα και στις περιπτώσεις αυτές όταν οι άνθρωποι ανώνυμα προβαίνουν σε ρητορική μίσους και θέλουν να επιτεθούν. Άλλωστε θα πρέπει να γίνει αναπερίπτωση έρευνα από την αστυνομία και να μην έχουμε απλώ ένα μαγικό φίλτρο που θα μπορεί να τους εντοπίσει όλους online. Αυτή είναι λάθος ιδέα. Ευχαριστούμε κύριο Μήλο. Um, what needs to be done? Τι πρέπει να γίνει. Το σημαντικότερο ερώτημα. Ο σκοπός και της επίσκεψής μας συζητήσαμε ενδελεχώς την κατάσταση αλλά προτείνω να έχουμε στεναρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις πλατφόρμες. Η απειλή του κανονισμού που ηγέρθη επανειλημμένος ίσως είναι το μόνο κίνητρο που οδήγησε τις πλατφόρμες να εφαρμόσουν πολιτικές ταχύτερα και αποτελεσματικότερα να κατεβάζουν αναρτήσεις με παρακίνηση σε μίσους. Υπάρχει το θέμα ισορροπίας ελευθερίας του λόγου, θεμητής παρέμβασης και ομιλίας, αλλά τώρα η νοοτροπία και η ζωή ανθρώπων καταστρέφεται σήμερα από λόγους μίσους, από ομιλίες μίσους, όπως είπαν οι συνάδελφοι. Πρέπει να δράσουμε. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι από ό,τι πριν. Να το παραλληλήσω με το GDPR. Εκ των πραγμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει προδιαγραφές για όλο τον κόσμο. Για την προστασία της ιδιωτικότητα, μοναδική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωση. μπορεί παρομοίως να κινηθεί και να καθορίσει προδιαγραφές για όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση δυνάμεων α, χειραγώγησης και παραπληροφόρησης. Αυτό που είπε ο κ. Γιούρικ. Ναι, Κάποια χρηματοδότηση παίρνουμε από τον Εθνικό Φορέα για τη Δημοκρατία μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από την κυβέρνηση παίρνουμε πόρους. Έχουμε πολλαπλούς πόρους χρηματοδότησης. Κύριε Ούρικ, εδώ εκπροσωπείται εδώ σε αυτό το βήμα πολιτικό κόμμα που συνέλεγε υπογραφές για δημοψήφισμα στην Σλοβακία για να αποχωρήσει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα απολαμβάνει τα ωφέλη εδώ ε, του να είναι ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πιο ενδιαφέρον είναι ένα συνάδελφός στο Κοινοβούλιο ε, καταδικάστηκε για παρακίνηση σε μίσος και απαγορεύτηκε η συμμετοχή του. Έπρεπε να παραιτηθεί το αξιώματό του του βουλευτού στο Κοινοβούλιο. Ε, λοιπόν, αυτό που να το λάβετε υπόψη. Γιατί σπήρει τον αντισημιτισμό και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Γιώρικ. Η κυρία Χιούγκεν ε, πάρα πολύ σύντομα γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά ήδη για τον κανονισμό, για την ομοθεσία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορεί να διαδραματίσει. Είναι γεγονός ορισμένες οργανώσεις μέλη μας συμμετέχουν στην κατάρτιση του κώδικα δεοντολογίας και στην παρακολούθησή του, αλλά εκφράζουμε κριτική για το ρόλο που παίζει δίνει συγχωροχάρτη στις πλατφόρμες και δεν τις μιλάει για ρύθμιση. Και επίση ποιο είναι ο ρόλο στο ΜΚΟ. Το σημαντικότερο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αναμένουμε εκείνοι που είναι εκτεθειμένοι στο μίσος ε, να δίνουν και αυτή τη λύση. Ορισμένοι υποστηρίζονται για να συμμετέχουν, άλλοι όχι. Τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμβαίνει παντού αυτό. Η κοινωνία των πολιτών έχει οργανώσεις που δεν υποστηρίζονται για να παίξουν το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην αντιμετώπιση του μίσου, στην υποστήριξη των θυμάτων και πολύ συχνά βλέπουμε χρήματα ε, τα, τα project να πηγαίνουν σε καινοτόμε λύσεις. Ενώ αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζονται οι οργανώσεις είναι υποστήριξη για την καθημερινή τους δουλειά που είναι πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ ανθεκτική. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε όταν μιλάμε στο πρόγραμμα ας πούμε, για τα δικαιώματα και τις αξίε. Πώ θα εξασφαλίσουμε τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας ε, σε ε, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ένωσης. Εκτός της Ένωσης έχουμε τέτοιο μηχανισμό, με τους δικούς μας τι κάνουμε. Βλέπω, Πρόεδρε, είστε έτοιμος να με σταματήσετε. Ένα τελευταίο, που ήταν πολύ σημαντικό επίσης, το μίσος Πολώνη. Και εγώ μιλώ εξ ονόματος κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, αλλά είναι ε, πρώτα μια μειονότητα που ε, ε, πλήττεται που βάλετε, μετά είναι η επόμενη και μετά η μεθεπόμενη. Είναι πολύ οριστηρό αυτό το έδαφος. Συνεργαζόμαστε για να δημιουργούμε συμμαχίες. Και τώρα, τέλος, χωρίς να γίνει διάλογος, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τα τρασφοβικά σχόλια να ακούγονται. Σέβομαι τις απόψεις όλων, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην μιλάμε εξ ονόματος άλλων ομάδων όπως ακούσαμε εδώ να γίνεται λόγος για φεμινίστριες, λεσβίες, γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Μπορεί να σέβομαι τη γνώμη σας και τη σέβομαι πολύ, αλλά προσοχή σας παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να μοιραστώ με όλους εσάς που απομείνατε εδώ ε, και στο πόντιουμ και στα έδρανα μερικά καταληκτικά σχόλια. Καλά κάνατε και ήρθατε εδώ. Η Επιτροπή μας νοιάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ε, συζητήσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Την κάνουμε αυτή τη συζήτηση τακτικά στην Ολομέλεια. Ασχολούμαστε με τα ζητήματα αυτά. Έχουμε κάνει εκθέσεις, έχουμε εγκρίνει εκθέσεις μέχρι τώρα και ψηφίσματα. Επίσης ξέρουμε ότι χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κράτους δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και δημοκρατίας που να ε, είναι συνολικό να συμπεριλαμβάνει όλους χωρίς διακρίσεις, χωρίς στιγματισμούς, χωρίς διαπόμβευση, χωρίς πολιτικά παιχνίδια και όπου κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάζεται σε τακτική βάση με ε, παραμέτρους αντικειμενικές. Στον ίδιο δρόμο που χαράξαμε όταν εγκρίναμε ε, το βαθμολόγιο για τη δικαιοσύνη, το περίφημο scoreboard. Και καλά κάνουμε και προσκαλούμε πάνελιστ για να μοιραστούν μαζί μας ε, τις εμπειρίες τους και την προσήλωση του μπορεί να συμφωνείτε με κάποιες από τις απόψεις αυτές και με άλλες να διαφωνείτε. Και καλά κάνετε. Ε, απλώς αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μας νοιάζει το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία και ιδιαίτερα αυτή η οπισθοδρόμηση. Αυτό το πισωγύρισμα και τα προβλήματα που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια από τότε που το έθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί υποτίθεται ότι αυτά είναι δεσμευτικά για όλους μας και μας θυμίζουν ότι ε, ε, οι αξίες του άρθρου 2 δεν είναι ευχολόγιο και ευσεβής πόθη, αλλά δεσμευτικά για όλους. Προστασία των μειονοτήτων, διάκριση των εξουσιών, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και το δικαίωμα των μειονοτήτων ε, να διαφωνούν με την κυβέρνηση και να φιλοδοξούν να γίνουν ε, ε, η μειοψηφία πλειοψηφία και η αντιπολίτευση συμπολίτευση. Το κράτος δικαίου δεν σημαίνει πάντα το κράτος του νόμου και δεν είναι η πλειοψηφία εκείνη που επιβάλλει το νόμο της. Δεν έχει το δικαίωμα η πλειονότητα να καταπιέζει τη μειονότητα και να την παρενοχλεί και να υπαγορεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ατομικά δικαιώματα κάθε πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά προστατεύονται από τον Ευρωπαϊκό ε, Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και καμία πλειοψηφία δεν έχει το δικαίωμα να κλονίζει τα ίδια τα θεμέλια μιας ένωσης που βασίζεται στο νόμο και υποτίθεται ότι εκεί κρατεί ο νόμος και το δίκαιο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, λοιπόν, καλά κάνατε και ήρθατε και τα είπατε εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους προηγούμενους τέσσερις. Ήταν πολύ εντατική ημέρα και συνεχίζεται αύριο στις 9 η ώρα ακριβώς. Καλό σας βράδυ και τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ.